Dear colleagues, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, που είναι η ακρόαση του υποψηφίου για, την, ε, για εκτελεστικό διευθυντή της ΕΜΑ και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μετά από την διαδικασία επιλογής ο κύριος Γκουιντοράτη επελέγει ως εκτελεστικός διευθυντής της ΕΜΑ. Στις 16 Νοεμβρίου 2011 για πέντε χρόνια αλλά υπήρξαν κάποια προβλήματα μέσα στα πέντε αυτά χρόνια και ξαναξεκινάμε τη διαδικασία διορισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, ΕΜΑ ξαναδιόρισε ως υποψήφιο τον κύριο Ράζη τον Οκτώβρη και οργανώνουμε αυτή την ακρόαση για να να θέσουμε ερωτήματα στον κύριο Ράζη και να εγκρίνουμε το διορισμό του. Δύο ώρες περίπου είναι, κρατάει η διαδικασία ακρόασης. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κύριο Ράζη να κάνει μια εισαγωγική παρέμβαση 10 λεπτών περίπου και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων. Ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση και στη συνεχεία 45 δευτερόλεπτα για συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό για την τελική απάντηση. Πρώτα απ' όλα θα δώσουμε τη δυνατότητα και μετά θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κύριο Ράζη να κάνει, να τα τελικά του σχόλια και μετά θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση της απόδοσης του κυρίου Ράζη σήμερα το απόγευμα στη συνάντηση των συντονιστών. Και ξεκινώ δίνω το λόγο στον κύριο Ράζη για την αρχική του ομιλία και μετά θα ξεκινήσουμε τις απαντήσεις και μετά τις ερωτήσεις. Thank you, Mr. Chairman. Members. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την ενθάρρυνση και για την υποστήριξη που μου έχετε παράσχει το προηγούμενο δύσκολο και μακρό έτος. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να είμαι ενώπιον σας σήμερα και να σας παρουσιάσω το όραμά μου για την ΕΜΑ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων και το σύστημα έγκρισης των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει τα μάλα. Νομίζω ότι περνάμε μια σημαντική μεταλλαγή στο σύστημα της ε, ανάπτυξης και έγκρισης φαρμακευτικών συσκευασμάτων η πιο μεγάλη αλλαγή που έχω δει στα 35 χρόνια της καριέρας μου στη δημόσια υγεία ως ιατρός, ερευνητής ή αρμόδιος για αριθμιστικές αρχές. Πιστεύω όμως ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας μπορούμε να περιμένουμε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες θα παρέχονται με τελείως διαφορετικό τρόπο όπως σήμερα. Τέσσερις λόγοι είναι για αυτή την αλλαγή. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια αυξανόμενη πολυπλοκότητα των φαρμάκων και επίσης αυξανόμενη πολυπλοκότητα της επιστήμης, των επιστημονικών γνώσεων που χρειάζονται για να προετοιμαστούν αυτά τα φάρμακα. Μετά από 40 χρόνια μοριακής βιολογίας έχουμε διαφορετικές πια ε, γνώσεις για την ε, προέλευση και τις αιτίες των ασθενειών ακόμα και σε μοριακό επίπεδο. Με αυτή την κατανόηση του πώς λειτουργούν τα φάρμακα σε αυτό το επίπεδο θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε νέα φάρμακα. Ένας δεύτερος λόγος είναι η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση της ανάπτυξης και παρασκευής φαρμάκων. Σήμερα πάνω από 85% από τα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία καταναλώνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τουλάχιστον ένα τμήμα της ε, διαδικασίας παραγωγής τους που λαμβάνει χώρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάνει την ε, αλυσίδα παραγωγής, αλυσίδα προμήθειας φαρμάκων ιδιαίτερα πολύπλοκη και ευάλωτη σε διαταράξεις. Οποιοδήποτε πρόβλημα παραγωγής σε οποιοδήποτε εργαστήριο στον κόσμο μπορεί να οδηγήσει σε μια ε, έλλειψη, σημαντική παγκόσμια έλλειψη σημαντικών φαρμάκων. Τρίτος λόγος είναι ο αριθμός και η πολυμορφία των εμπλεκομένων για την ε, παροχή φαρμάκων στους ασθενείς από το επίπεδο των αρχικών εργαστηριακών δοκιμών μέχρι να συνταγογραφηθεί ένα φάρμακο. Για πολλά χρόνια η ρύθμιση για τα φαρμακευτικά σκευάσματα έχει γίνει με έναν τρόπο απομονωμένο. Σήμερα όμως οι ρυθμιστές πρέπει να εργαστούν με πολλούς εμπλεκομένους σε αυτή τη διαδικασία, με τους ερευνητέ, με τις εταιρείες, τους επενδυτές, τα σώματα αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας, με ασθενείς και με τους ε, εργαζόμενοι στον υγειονομικό τομέα. Συνεργαζόμαστε ήδη με πολλούς από αυτούς, αλλά ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε από την απλή συνεργασία στην πλήρη ολοκλήρωση για να μπορούν τα φάρμακα να φτάνουν πιο γρήγορα στους ασθενείς. Τέλος, υπάρχει ένα τέταρτο στοιχείο που είναι ότι η νομοθεσία που εσείς εγκρίνετε παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Πρόσφατα η νομοθεσία φαρμακο επαγρύπνησης έχει τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε και ρυθμίζουμε την ασφάλεια των φαρμάκων στην Ευρώπη. Ακόμα πιο πρόσφατα, ο κανονισμός για τις κλινικές δοκιμές που έχει εισαγάγει το πιο διάφανο σύστημα έγκρισης, εποπτείας και παράδοσης αναφορών για τις κλινικές μελέτες. Και επίσης έχουμε την νομοθεσία την, στον ε, κτηνιατρικό τομέα που ελπίζουμε ότι θα φέρει πιο καινοτόμα φάρμακα για τα ζώα. Γενικά, αυτοί οι κανόνε έχουν βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα τη αξιολόγησή μα για τα φαρμακευτικά συσκευάσματα, αλλά έχουν προσθέσει συγχρόνω και περισσότερη πολυπλοκότητα στι διαδικασίε μα. Αναφέρομαι λοιπόν για μια μεταλλαγή, για μια μεταμόρφωση, η οποία έχει μεγάλο δυναμικό για να ε, ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ασθενών στην Ευρώπη. Όλοι θέλουμε να έχουμε μια τέτοια αλλαγή Πρέπει όμως να καθοδηγήσουμε αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι και οι προκλήσεις ώστε αυτό το οποίο θα γίνει σε τελική ανάλυση θα είναι προς το όφελος των ασθενών στην Ευρώπη. Ένα λοιπόν από τα βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα της βιωσιμότητας και βλέπω τρία επίπεδα στα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της βιωσιμότητας. Πρώτα απ' όλα η βιωσιμότητα των συστημάτων μας για υγειονομική περίθαλψη. Τα νέα φάρμακα μπορούν να δημιουργήσουν νέες συνθήκε σε πολλά υγειονομικά συστήματα της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να επωφεληθούν πολλοί ασθενείς από την τεράστια επιστημονική πρόοδο που έχουμε κάνει τα τελευταία 40 χρόνια. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η βιωσιμότητα του δικτύου κανονισμών για τα φάρμακα στην Ευρώπη. Είναι τόσο μεγάλη πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουμε που οι ρυθμιστές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες πρώτης τάξεως. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη να προσφεύγουμε σε όλο και πιο εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Οι εθνικές αρχές λοιπόν και η ΕΜΑ θα πρέπει να μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Τρίτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα τη έρευνα και τη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το κόστο τη έρευνας αυξάνεται, ενώ συγχρόνω δεν έχουμε τι επενδύσει για την ανάπτυξη περαιτέρω φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κέρια η έρευνα και η ανάπτυξη, όχι μόνο για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα, αλλά κυρίω για να έχουμε καλύτερε θεραπείε για του ασθενεί. Αυτό περιλαμβάνει και τι ε, ε αναδιόμενες ασθένειες όπως η έμπολα, αλλά και τους παλιούς εχθρούς που μπορεί να επανέλθουν. Και εδώ υπάρχει το θέμα της αντιμικροβιακής αντίστασης και την ε, έλλειψη φαρμάκων για να αντιμετωπίσουν μολύνσεις από βακτηρίδια τα οποία έχουν πολλαπλή ανθεκτικότητα. Πώ θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν όλε αυτέ τι ε, προκλήσει. Όταν ξεκίνησα στην ΕΜΑ το 2011, είχα ένα σαφέ θεματολόγιο. Πρώτα απ' όλα να έχουμε μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με το να αλλάξουμε τι δομέ τη ΕΜΑ και να προσαρμόσουμε τις διαδικασίες στον χρόνο ζωής των φαρμάκων. Δεύτερον, να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους εμπλεκόμενους και από το κοινό για το έργο του φορέα μας. Παραδείγματο χάρη η πολιτική μα σε σχέση με τη δημοσίευση των στοιχείων κλινικών ε, μελετών και οι δηλώσει ε, συμφερόντων για να εξασφαλίσουμε ότι υπήρξε σωστή διαχείριση των αντιμαχωμένων συμφερόντων και πρόσβαση στην καλύτερη εμπειρογνωμοσύνη. Εγώ θέλω και είμαι δεσμευμένο να συνεχίσω τον αγώνα για μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα τη ανάπτυξη φαρμάκων και τη αξιολόγηση. γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η θεμέλη για την εμπιστοσύνη του κοινού στο έργο μα για το καλό όλων. Επίση πρέπει να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα. Πρέπει να μειώσουμε το χρόνο που χρειάζεται για την έγκριση ενός φαρμάκου με, από την έγκριση μάλλον φαρμάκου μέχρι την διαθεσιμότητά του για τους ασθενείς. Συγχρόνως όμως πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα νέα και τόμα φάρμακα είναι ασφαλή. Αυτό σημαίνει πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ε, προβλεψιμότητα των διαδικασιών μας για αυτούς που αναπτύσσουν νέα φάρμακα, συγχρόνως όμως να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τα σώματα αξιολόγηση υψηλής τεχνολογίας ώστε να μπορεί να γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία αποφάσεων και έγκρισης. Τα νέα εργαλεία λοιπόν τα οποία έχουμε τώρα με την νομοθεσία περί, περί φάρμακο επαγρύπνησης μας επιτρέπουν να καταλάβουμε καλύτερα ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος των φαρμάκων στο καθημερινό επίπεδο και πώς χρησιμοποιούνται στην πράξη. Στην Ευρώπη έχουμε ένα πληθυσμό 500 εκατομμυρίων πολιτών και γι' αυτό έχουμε πολλές ευκαιρίες να εξετάσουμε και την ασφάλεια αλλά και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Είναι λοιπόν ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Αυτά είναι λοιπόν κάποιες από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων και κάποια από, τα, από τους δρόμους και από τις λύσεις που θα βοηθήσουν την βιωσιμότητα του συστήματος και την ποιότητα των αξιολογησεών μας. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με αποτελεσματικό τρόπο αν συνεργαστούμε από κοινού όλοι οι εμπλεκόμενοι και φυσικά θα πρέπει να έχουμε την δική σας βοήθεια. Χρειαζόμαστε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, χρειαζόμαστε το Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση στο όλο θέμα των φαρμάκων καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, ώστε να έχουμε πραγματική βελτίωση και καινοτομία στην υγειονομική περίθαλψη να βοηθήσουμε λοιπόν να, σας ασθενείς να βελτιώσουν τη ζωή τους με ένα κόστος το οποίο είναι προσιτό στην κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Uh, our... Ευχαριστώ και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε, λέει ο Πρόεδρος, τον πρώτο γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές. Ένα λεπτό για το ερώτημα, δύο για τις απαντήσεις, 45 δευτερόλεπτα για την ε, Επόμενη για συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό για την απάντηση. Ο Πέτερ Λίζε είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε καλή εμπειρία μαζί σου και νομίζω ότι ξέρουμε ότι είσαι έτοιμος να συγκεντρώσεις πάντα την προσοχή σου στα θέματα αυτά. Ως μικροβιολόγος θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο έφτιαξες που είναι το θέμα της ε, αντιμικροβιακής αντίστασης και ξέρουμε ότι υπάρχει μια πρόταση της Κομισιόν για νέα αντιβιωτικά για τα ζώα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των νέων αντιβιωτικών για τους ανθρώπους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να υποστηρίξει την πρόταση της Κομισιόν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό σε μια ειδική πρόταση της Κομισιόν για το πώς θα μπορέσουν τα καινοτόμα φάρμακα για τους ανθρώπους να έρθουν στην αγορά, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν τις κατάλληλες συνθήκες πλαισίου για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να ξέρω τι μπορεί να κάνει η αίμα για να βοηθήσει αυτή την κίνηση. Κύριε Λίζο, ευχαριστώ για την ερώτησή σα, Λέει ο κύριο Ράζη. Νομίζω ότι θίξατε έναν από τους τρεις πυλώνες τη δυνατότητα να έχουμε νέα αντιβιωτικά και νέα εργαλεία για αυτά τα τόσο ανθεκτικά βακτηρίδια. Και ακριβώ αυτό ο άξονα με απασχολεί, αυτό ο πυλώνα δηλαδή, η ρυθμιστική πλευρά του θέματος, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχουμε συγκροτήσει αυτή την ε, task force η οποία παγίως ασχολείται με το τι μπορούμε να κάνουμε με τα μέσα που έχουμε στα χέρια μας και κατά πόσο μπορούμε να προτείνουμε κάποια καινούργια εργαλεία ούτως ώστε να μπορέσουμε να διευκολυνθούμε και να έχουμε κάποιο είδους ε, συνοπτική ταχεία διαδικασία σε σχέση με τα αντιβιωτικά που θα έχουμε. Πρόκειται για πολύ σημαντικό κομμάτι του όλου συστήματος. Οπότε δε άπαξ και λάβαμε αυτή την τοποθέτηση και είναι και θέμα επιστήμης. Είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια μέτρα ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα νέα φάρμακα, τα νέα αντιβιωτικά, ούτως ώστε να δούμε κατά πόσο θα συνταγογραφούνται ορθώς και τα τυχόν ε, αντιβιωτικά να μην διατρέχουν τους ε, κινδύνους τους σημερινούς. Δηλαδή το να προκαλούν ε, ανθεκτικότητα. Οπότε γι' αυτό και πιστεύω ότι έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα μέσα ούτως ώστε να μπορούμε να παράσχουμε συμβουλές στις εταιρείες να παραγάγουν αυτά τα φάρμακα αλλά όπως έλεγα πρόκειται για ολιστική προσέγγιση. Να δούμε τι θα γίνει με μακροπρόθεσμα, κατά πόσο θα μπορέσουμε να έχουμε το κατάλληλο περιβάλλον, τόσο ώστε να διεκπεριώσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Λίζε. Θα ήθελα κάτι πιο συγκεκριμένο, αν μπορείτε. Χρειαζόμαστε νομικό πλαίσιο, πιστεύω, το οποίο εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις για τα νέα φάρμακα γιατί φυσικά απαιτούν μεγάλες επενδύσεις και δεύτερον τα νέα φάρμακα να μην είναι η πρώτη επιλογή μέχρι ότου δοκιμαστούν σωστά. Ένα σύστημα λοιπόν το οποίο δίνει κίνητρα στην Κομισιόν αλλά δεν οδηγεί και σε μεγάλο κόστος για αυτούς. Θα ήθελα λοιπόν να έχω τη δική σας άποψη για το πώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια πρόταση Κομισιόν η οποία εξασφαλίζει αυτό το στόχο. Ε, thank you for, for... Ευχαριστώ για αυτά που διευκρινίσατε. Όντως, θα έπρεπε να υποστηρίξουμε και θα υποστηρίξουμε την ε, τελική πρόταση. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, ούτω ώστε να είναι τεχνικά βιώσιμη μια τέτοια προσέγγιση, ούτω ώστε επίσης να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε, να υποστηρίξουμε αυτές τις επενδύσει. γιατί γνωρίζουμε ότι τα περιθώρια που υπάρχουν είναι στενά, όμως βρισκόμαστε στην ε, πορεία του να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Είμαστε σε ετοιμότητα. Thank you now, Matthias vielen Dank. Ο Ματίας Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράζη. Ως αρμόδιος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ΕΜΑ θέλω να σε ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε το 2011 και την εποχή που ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος είχαμε μια πολύ καλή και ε, μέσα στα πλαίσια διαφάνεια συνεργασία μαζί σας. Για τη δική μας πολιτική ομάδα τώρα, η πρόσβαση στα φάρμακα στις υγειονομικές ε, υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί είναι πολλά κράτη-μέλη ξεχνούν ότι δεν βρισκόμαστε πριν από 10 ή πριν από 15 χρόνια. Αυτό ήταν σαφές από αυτά που είπες ότι όλος ο τομέας υγειονομικής παρε... πα... παροχής υπηρεσιών έχει αλλάξει άρδιν. Εμείς ε, είχαμε οργανώσει μια task force, είχαμε κάνει μια ακρόαση για τα θέματα αυτά και από την ακρόαση αυτή προέκυψε ότι όλος ο τομέας των ε, ε, αξιολογήσεων υψηλής τεχνολογίας είναι κέριος. Και η Κομισιόν και η ΕΜΑ λοιπόν έχουν υποσχεθεί ότι θα υπάρξει βελτίωση στο σύστημα αυτό. Από τη δική σας πλευρά λοιπόν, από την πλευρά της ΕΜΑ, τι προβλέπετε να γίνει και για το θέμα αυτό των αξιολογήσεων και εμείς τι μπορούμε να περιμένουμε από τη δική σας πλευρά. Γιατί για μένα η διαδικασία αυτή αξιολογήσεων είναι κέρια για να μπορούμε να έχουμε σωστές υπηρεσίες υγειονομικού χαρακτήρα αλλά και ανάπτυξη νέων φαρμάκων τα οποία θα είναι και ε, προσιτά στους ασθενείς. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας κύριε Γκρότ. Η δέσμευσή μας ως υπεύθυνη για την αξιολόγηση είναι όταν η ΕΜΑ δώσει την αδειοδότηση να δούμε για την διάθεση στην αγορά πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό Αυτή η αδειοδότηση για τα φάρμακα είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να δούμε εμείς πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ως αίμα. Ως υπεύθυνοι για την τεχνολογική αξιολόγηση έχουμε να κάνουμε με 60 συμβουλές για τέτοια προϊόντα. Είναι δύσκολο να συνεργαστούμε ως δύο διαφορετικές κοινότητες, αλλά ξέρουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Στο μέλλον, για να προωθήσουμε την καινοτομία και για να είναι προσβάσιμη και στους ασθενείς, θα πρέπει ευθύ εξ αρχής να ακολουθήσουμε δύο διαδικασίες, από όσον βλέπω. Πράγμα που θα είναι επωφελές για τους ασθενείς, διότι ο ασθενής δεν θα υφίσταται πολλές νέες δοκιμές. Θα είναι τα θέματα πιο απλά και θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία αξιολόγησης. Θα έχουμε λιγότερες δοκιμές και πιο εύκολη και ταχεία πρόσβαση των ασθενών. Εάν συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και βελτιωθεί, θα είναι θετικό αυτό, αλλά όπως είπα και στην αρχική μου παρατήρηση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε την ε, συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο κοινοτήτων με καλύτερο τρόπο. Ε, ευχαριστώ, λέει ο Γκρότε. Συμπληρωματικό ερώτημα. Είναι σίγουρο ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Τι θα περιμένατε όμως τότε εσείς από το Κοινοβούλιο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των ε, τεχνολογιών, τεχνολογικών αξιολογήσεων υψηλού επίπεδου. Είναι θέμα καλύτερης χρηματοδότησης, είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε στον προϋπολογισμό και εδώ είναι παρόν ο νέος Γενικός Διευθυντής ε, της Κομισιόν. Καλώς ήλθατε. Ίσως και αυτός μπορεί να μας διαφωτίσει περισσότερο. Αν υπάρχουν ε, λοιπόν νέες ε, ενέργειες θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν και την κατάλληλη χρηματοδότηση. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα πληρώνει κιόλα όταν υπάρχει η έγκριση νέων φαρμάκων, τι τέλη θα πρέπει να επιβάλλονται και σε ποιους. Αλλά το ερώτημα μου και πάλι είναι να μάθω πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει ώστε να επιτευχθούν όλα αυτά. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ το χρόνο και να σας απαντήσω σύντομα. Αυτό το οποίο ζητώ είναι υποστήριξη της κοινή δράσης μεταξύ ΕΜΑ και Κομισιό για την ενίσχυση και προώθηση αυτών που προβλέπεται. Θα έχουμε δηλαδή την, θέλουμε την κατάλληλη νομοθεσία και θέλουμε τους κατάλληλους πόρους δεν ζητούμε περισσότερα από ό,τι χρειαζόμαστε, αλλά αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια νέα δραστηριότητα, θα πρέπει να μπορούμε να την προωθήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο και να έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται. Thank you very much. And now for uh, Mr. Pieka for the e Dziękuję panie przewodniczący, panie profesorze. <clears throat> zajmę się... Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω στην διαδικασία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για την αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών συσκευασμάτων και επίσης για την ασφάλειά τους σε ό,τι αφορά τον ασθενή. Εδώ έχω ένα ουσιαστικό για μένα ερώτημα. Η διαδικασία έγκρισης ε, στην αίμα είναι μια μακροσκελής διαδικασία ενώ σήμερα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις, ιδίως όπως ελέγχθη για τα αντιβιωτικά, για τα ογκολογικά θέματα, για τις σπάνιες ασθένειες. Και για αυτές τις προκλήσεις έχει αναπτύξει ο φορέας σας κάποια σχέδια για το πώς μπορεί να προχωρήσει με τα θέματα αυτά. Προσπαθείτε να έχετε μια αναδιάθρωση τις, ε, τις υπηρεσίες σας ώστε να γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία έγκρισης και θα μπορούν έτσι τα κοινοτόμα φάρμακα να εγκρίνονται πιο γρήγορα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε την κατάσταση μιας ε, κεντρικής διαδικασίας για ορισμένα φάρμακα βιολογικού χαρακτήρα. Εσείς υποστηρίζετε την κεντρική διαδικασία ή ή αποκεντρωμένες. Thank you, Mr. Well, I think... Uh, Νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δύο ε, ε, πρωτοβουλίες ώστε να διευκολυνθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική η όλη διαδικασία και λιγότερο χρονοβόρα. Η πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πρωτοβουλία STAMP ώστε να υπάρχει ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε νέα φάρμακα και έχουμε και μία ε, πιλωτική πρωτοβουλία ώστε να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε τα υποσχόμενα για το μέλλον φάρμακα τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε καθ' όλη τη διάρκεια της Ανάπτυξη τους και προσπαθούμε με την τρέχουσα νομοθεσία να προωθήσουμε και μια άλλη πρωτοβουλία, την Τραπράιν, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίζουμε και τα υποσχόμενα φάρμακα που έρχονται από τη Σμιμία όπου δεν υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ε, γνώση και ίσως και πόρη για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν μόνες τους όλη την διαδικασία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι στην ΕΜΑ μπορούμε με αποτελεσματικό τρόπο να υποστηρίξουμε και να οδηγήσουμε ε, τις ε, επιχειρήσεις αυτές ώστε να χρησιμοποιήσουν με το καλύτερο τρόπο τους πόρους που διαθέτουν και, για... και πολλές φορές να τους οδηγήσουμε στο να περικόψουν τις διάφορες δραστηριότητες οι οποίες ίσως δεν χρειάζονται για να τους ενισχύσουμε στις γνώσεις που πρέπει να έχουν για να λάβουν δραστηριότητες πολύπλοκες. Έχετε λοιπόν την άποψη ότι χρειάζονται νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να μπορούν να έρχονται τα φάρμακα πιο γρήγορα στην αγορά. Και άλλο ένα ερώτημα το οποίο είναι σημαντικό αλλά ίσως δύσκολο είναι έτοιμη, είναι έτοιμη η αίμα να προχωρήσει σε μία μορφή... Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν ακούγεται η μετάφραση. Είναι έτοιμη να προχωρήσει σε φιλελευθερωποίηση. Może jeszcze raz. No, chodzi switch to the English. Yes. Για να ακούσω τρόπο τα αγγλικά. Okay. Is okay? Okay. Chodzi mi o usprawnienie procesu rejestracji i czy σε σχέση με αυτήν την ε, διαδικασία της καταχώρησης στο Μητρό. Θα πρέπει να πρετανεύει η διαφάνεια ή σε αυτές τις κλινικές δοκιμές και αυτό θα πρέπει να γίνει γρήγορα διότι το νέο αντιβιωτικό θα πρέπει να είναι έτοιμο να χορηγηθεί στους ασθενείς. Οπότε θα πρέπει εδώ να εξετάσουμε το θέμα της ε, ε, ανθεκτικότητας και της αντοχής στους μικροοργανισμούς. Uh, yes, certainly. Ναι, βεβαίως λέει κύριε Ράζη. Βεβαίως και θα πρέπει να βελτιώσουμε την νομοθεσία ούτω ώστε να διεκπεριώνουμε ταχύτερα την διαδικασία για το θέμα το οποίο εσείς θίξατε. Βεβαίω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως νομίζω ότι στην ισχύουσα νομοθεσία έχουμε πολλές λύσεις που δεν όμως και τόσο ε, αυστηρές. Οπότε γι' αυτό και ε, η αίσθησή μου θα πρέπει ό,τι έχουμε το χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Οπότε και να δούμε κατόπιν πώς θα πρέπει να κάνουμε τις μικροαλλαγές που χρειάζεται η κείμενη νομοθεσία. Ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Και μην κάτσουμε από το α να φτιάξουμε νέα νομοθεσία. Thank you very much. And now, Madame Merci, Monsieur le Président. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλώ ορίσατε. Και θα ήθελα να χαιρετήσω και τον κύριο Νίστικο, τον πρώην συναδελφό σα, με τον οποίο βιαστήκαμε για διάφορα προβλήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολλά ελέγχθησαν ήδη και ξέρω ότι έχουμε λίγο χρόνο. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπατε για την διαφάνεια. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για μας, για τους Ευρωπαίους πολίτες το θέμα αυτό και υπενθυμίσατε ότι το 2011 ήταν ο κύριος άξονας της ε, δραστηριοτήτους. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να μιλήσω για τα θέματα που αφανούν τη δημοσίευση των δεδομένων των φαρμακευτικών εταιριών. Είπατε ότι το σύστημά μας είναι το πιο διαφανές και είπατε ότι θέλετε να δημιουργήσετε κινήτρο ώστε να, να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια. Στην ε, πράξη τι σημαίνει για σας αυτό, περισσότερη διαφάνεια, κυρίως όταν υπάρχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για τους πολίτες που μας ακούν και μας βλέπουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου με επαναφέρετε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Περισσότερη διαφάνεια. Νομίζω ότι είμαστε στο προβλέπουμε τη διαφάνεια σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε ήδη διάφορους συναδέλφους σε άλλα μέρη του κόσμου που κάπως ε, εκνευρίζονται από αυτή την... Ότι πάλι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την διερμηνία. Έχει χαλάσει το μικρόφωνο, κάποιο μικρόφωνο χαλασμένο στη γερμανική καμπίνα, λέει ο κ. Γκρότ. <clears throat> δεν, γιατί δεν ακούμε τίποτα. Okay. Okay. You can continue. Yeah. Ε, So, uh, for the clinical uh, um, data, Για τα ε, δεδο... κλινικά δεδομένα. Όταν αρχίσουμε, θα αρχίσουμε να διαθέτουμε στοιχεία και θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα. Καλό είναι να έχει κανείς ε, δεδομένα και να τα χρησιμοποιεί όμως με ευφυή τρόπο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει στο χρόνο να το βελτιώσουμε. Η τεχνολογία βεβαίως θα μας βοηθήσει στο μέλλον να κάνουμε τη δουλειά μας ε, καλύτερα. Τώρα όσον αφορά τα επληκόμενα συμφέροντα, δεν είμαστε αστυνομική αρχή. Πρέπει να επαφιέμαι σε κάποια στοιχεία που μας δίνουν, αλλά πρέπει να είμαστε πιο προσεκτική, να κάνουμε κάτι περισσότερο. Και βεβαίως ε, θα πρέπει αν υπάρχει πρόβλημα τέτοιου είδους συμφερόντων να μας τα επισημαίνουν κάποιοι, γιατί όπως σας είπα δεν είμαστε αστυνομική αρχή. Αλλά βεβαίως δεν μπορούμε πάντα να βασιζόμαστε σε ό,τι έχει λεχθεί από κάποιον. Δεν υπάρχει αυτό. Και βεβαίως χρειαζόμαστε εδώ και θεσμική υποστήριξη και κανόνες εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από ό,τι σήμερα στον τομέα αυτό. Επίσης μας απασχολούν ε, κάποιοι περιορισμοί που έχουμε εξαιτίας των ε, πόρων που διαθέτουμε, διότι έχουμε γύρω στους 30.000 πραγματογνώμες στο σύντομο το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Διαβάζοντας και πάλι το εξαιρετικό και εντυπωσιακό βιογραφικό σας, μας εντυπωσιάζουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως το γεγονός ότι την αρχή της σταδιαδρομίας σας ε, είχατε ε, σχέσεις με τους ε, εταίρους Αμερικανούς, με την FDA, όσον, γιατί... Τώρα, όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές της FDA, που σας ε, φαίνονται οι καλύτερες και τις οποίες εμπνεόμαστε, χωρίς ε, εδώ να μιλήσω για το πρόβλημα που υπάρχει με το TTIP, πώς βλέπετε την ενίσχυση των ε, διατλαντικών σχέσεων με μας και κυρίως το θέμα της πρόσβασης σε φάρμακα ασθενών που ε, πάσχουν από αυτό το οποίο ονομάζεται μία σπάνια ασθένεια και χρειάζεται γι' αυτό το λόγο να αντιμετωπιστεί τέτοιου είδου ασθένειε αποτελεσματικά να γίνουν περισσότερη έρευνα και στην ε, Ευρώπη από τους επιστήμονες. Εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα σε καμία σχέση με το TTIP. Για αυτά τα φάρμακα προβλέπονται για τις σπάνιες και ως φανές ασθένειες όπως λέγεται. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα σε αυτά, η πολιτική διαφάνεια που ακολουθούμε. Αυτό που ζητώ και κάνω έκκληση είναι να μην αμβληθεί ότι έχει γίνει ήδη για λόγους διαφάνειας σε θέματα δοκιμών για τέτοιου είδους φάρμακα. Προσπαθούμε με την FATPAC, με την Pride να έχουμε μία καλύτερη προσέγγιση και να υποστηρίξουμε ότι έχει γίνει ήδη στον τομέα αυτό. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για τους Ευρωπαίους πολίτες και ιδίως για το κόμμα μου η υγειονομική περίθαλψη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα φάρμακα ε, εξελίσσονται με έναν τρόπο ο είναι αντικειμενικός και προστατεύει την υγεία των πολιτών και επίσης και το κρατικό τον κρατικό προϋπολογισμό, ότι δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά. Θέλουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε ε, ολίσθηση μέσα σε εισαγωγικά στα θέματα αυτά. Ξέρουμε ότι υπήρξαν πάρα πολλέ ε, κριτικές που έχουν διατυπωθεί εναντίον των φαρμακευτικών εταιριών σε ό,τι αφορά την έλλειψη διαφάνεια στην διαδικασία ανάπτυξη νέων φαρμάκων για τι ε, ενδεχόμενε συγκρούσει συμφερόντων κτλ η ΕΜΑ παίρνει τα 83% του προϋπολογισμού της από ιδιωτικούς φορείς, από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πώς επιτρέπεται λοιπόν να ληφθούν υπόψη και τα συμφέροντα του ιατρικού τομέα ενώ συγχρόνως είσαστε ε, υπό την πίεση των λόμπι των επιχειρήσεων. Κάπου θα πρέπει να υπάρξει μια ε, οριοθετική γραμμή. Επίσης θα υπάρξει το θέμα τη τίζα της συμφωνίας αυτής. Θεωρείτε ότι μια τέτοια συμφωνία οδηγεί σε θετικέ ή αρνητικέ εξελίξει. Σα ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σα. Και πάλι. Και αυτό είναι ένα από τα κέρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα. Είναι γεγονό ότι πάνω από 80% του εισοδήματό μα έρχεται από τέλη που εισπράττουμε από φαρμακευτικές εταιρείες. Πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι παρέχουμε μια υπηρεσία και δεν τους δίνουμε κάτι δωρεάν. Γενικά, οι φαρμακοβιομηχανίες είναι ικανοποιημένες αν δώσουμε μια ακριβοδίκαια αξιολόγηση γιατί τους ικανοποιεί και έναντι των ανταγωνιστών τους. Γι' αυτό χαίρονται όταν είμαστε αυστηροί, αλλά πρέπει να είμαστε συνεπείς και συνεκτικοί σε αυτά που κάνουμε. Η συνεκτικότητα και η ε, αυστηρότητα σε ό,τι αφορά το επιστημονικό έργο είναι τα κλειδιά για να μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι και έναντι του κοινού και έναντι αυτών οι οποίοι περιμένουν κάποια υπηρεσία από εμά, δηλαδή τον φαρμακο... φαρμακευτικό τομέα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα ε, καλύτερης ε, διαφάνειας και εδώ απαντώ στο προηγούμενο ερώτημα. Αν μπορεί λοιπόν η, η φαρμακοβιομηχανία να διευκολύνει το δικό μας έργο ώστε να εξασφαλίσει και την απόσταση που πρέπει να έχουμε από αυτούς και τη διαφάνεια. Επίσης τον έχουμε μια επιτροπή επιπλέον. Αυτό μπορεί να <clears throat> οδηγήσει σε ε, Αλλά Τώρα έχουμε μια επιτροπή που έρχεται από 20, χρο... από 20 κράτη μέλη. Με την εμπειρογνωμοσύνη τους θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερη απόσταση από τα συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία εμπλέκονται. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω ένα συμπληρωματικό ερώτημα για τα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών. Σας ζήτησα να λάβετε κάποια θέση για τα θέματα αυτά και υπάρχει επίσης και η Συμφωνία Τίζα που παίζουν σημαντικό ρόλο τα φάρμακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως θα έχει μια απόσταση σε σχέση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα Εγώ δεν είμαι σίγουρος για την ανεξαρτησία που έχετε εσείς όμως ως φορέας. Να σας πω, Ζάζη, οφείλω να παραδεχθώ ότι δεν είμαι και τόσο εξοικειωμένος με το κείμενο στο οποίο παραπέμπεται. Πάντω θεωρώ ότι αν θεσπίσει κάποιου κοινού κανόνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι, συμπαθάτε με, έκανα λάθο τότε αυτό θα πρόκειται για κάποια δόκιμη πρακτική και εμείς θα ακολουθήσουμε. Πάντως στην υπηρεσία μας έχουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει να υιοθετούμε συγκεκριμένα μέτρα. Σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε πάντως, εγώ θα ε, εξήθαζα για το κατά πόσον όλα αυτά συνάδουν προς το στόχο μας. Δηλαδή να είμαστε προσεκτικοί και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε που να συνέβη προς το, τα όσα ισχύουν για να μην ανατρέψουμε όλα όσα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Κυρία Ριβαζή για τους Πρασίνους. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίσατε κύριε κιουτοράζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση για τη νανοστοιχεία. Ε, ε, Νονοσωματίδια. Λέει η κυρία Μπάκοσκα ότι θα πρέπει τα νανοσωματίδια να απαγορευτούν στα καλλιντικά. Το ψηφίσαμε στο κοινοτική κυρίως όσον αφορά της διοξινής τιτανίου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η απαγόρευση για λόγους ε, υγείας δεδομένου ότι εισχωρούν αυτές, ε, αυτά τα σωματίδια στο ε, σώμα Ο, υπέροχο, ο, υπέ, υπεύθυνος επίτροπος να μας λέει ότι δεν μπορώ να σας δώσω τον ε, λεπτομεριακό κατάλογο τέτοιου είδους νανοσωματιδίων που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Απ' την άλλη μία λοιπόν δεν έχουμε καταχώρηση σε επίπεδο φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τα εμβόλια και τα νοσοματίδια που χρησιμοποιούνται. Εσείς ε, αναλαμβάνετε τη δέσμευση να κάνετε αυτό το, ε, αυτή την εργασία καταχώρησης όλων αυτών των ανασωματιδίων. Αυτά τα ανανοσωματίδια δεν έχουν την ίδια, δεν είναι τα ίδια με τα υπόλοιπα σωματίδια. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Thank you for this challenging question. Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, πρόκληση. Μπορώ να σας πω ότι εμείς δεν θα με τα καλλιντικά. Για τα φαρμακευτικά προϊόντα ακόμη δεν έχουμε κατάλογο των ανασωματιδίων. μπορούμε να έρθουμε σε επαφή περισσότερο με άλλους οργανισμούς, την EDICOM, την ΕΚΑ, την ECBC, που ίσως θα είναι σε θέση να μας διευκολύνουν για να έχουμε στη διάθεσή μας αυτό τον κατάλογο. Μπορούμε να εστιάσουμε και εκεί την προσοχή μας. Εάν υπάρχει κίνδυνο στα φαρμακευτικά προϊόντα για εξαιτίας της ποσότητας τέτοιου είδους σωματιδίων που συμπεριλαμβάνονται σε σχέση με την περιοκτικότητα που υπάρχει ίσως και σε άλλα προϊόντα και ίσως η πολύ μικρή ποσότητα στα φάρμακα είναι πολύ ε, λιγότερη από ότι όταν χρησιμοποιούνται ανασωματίδια σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες σε άλλα προϊόντα. Ελπίζω λοιπόν ότι όσο πιο γρήγορα ε, ξέρουμε περί τίνος πρόκειται με τα νανοσωματίδια αυτά, τώρα καλύτερα θα είναι τα πράγματα στο μέλλον για τα φάρμακα. Σε 30 δευτερόλεπτα. Είστε συνομιλητής κλειδί, δεδομένου ότι εσείς δίνετε τις εγκρίσεις για τα φάρμακα στην αγορά. Μπορούμε να έχουμε σε κάθε φάρμακο με διαφάνεια ε, τις ενδείξεις για τα νανοσωματίδια που χρησιμοποιούνται είτε καθάνονται και μετά θα πρέπει να γίνει μια ειδική αξιολόγηση δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οι ίδιες ιδιότητες χημικές και φυσικές για το καθένα από αυτά. Σωστά. Δεν, υπάρχουν, δεν έχουμε τις ίδιες ιδιότητες. Δεν έχουμε όμως από όσο γνωρίζω, νομική βάση που μας επιτρέπει να επιβάλλουμε να χορηγούνται από τώρα τέτοιου είδους πληροφορίες. Πιστεύω παρά αυτά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το μελετήσουμε το θέμα αυτό, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να δούμε πού υπάρχουν σε κάθε προϊόν τέτοιου είδους νάνο σωματίδια. Δεν είναι προς το παρόν νομίζω θέμα δημόσιας υγείας, αλλά ίσως στο μέλλον θα δημιουργηθεί πρόβλημα και συμφωνώ μαζί σας όσο πιο ενωρίς ξεκινήσουμε τις διαδικασίες τόσο καλύτερα θα ε, καλύψουμε την κατάσταση και θα αποφύγουμε του κινδύνου εκ μέρου ε, ε, από τη χρησιμοποίηση τέτοιων νοσοματιδίων στο μέλλον. Ευχαριστώ. Είμαι πρόεδρε και καθηγητά Ράζη. Επί τη βάση προσφάτων μελετών, τι γίνεται όσον αφορά αυτά τα γενώσιμα. Λέει κάποια μελέτη ότι μέσα σε μία δεκαετία περίπου είναι δυνατόν να έχουμε εξοικονόμηση από 12 μέχρι 33 δις. Τι λέτε, τι δική σας υπηρεσία ούτως ώστε να είναι πιο εύκολη πρόσβαση στα αυτά γενώσιμα και τα συναφή γιατί επίσης έχει παρατηρηθεί ότι οι φαρμακοβιομηχανίες κατά 90% έχουν κάποιες ενεργές ουσίες που σπονθεύονται από την Κίνα και για αυτές τις ουσίες τι γίνεται έχουμε κακή διαχείριση των ε, απορριμμάτων και αποβλήτων οπότε μολύνονται πάρα πολύ τα ύδατα οπότε γίνεται ακόμα χειρότερη η αντοχή των μικροβίων. Άρα δεν θα πρέπει να δείτε τι γίνεται, από πού προέρχονται αυτές οι ουσίες. Άρα, τι πρέπει να κάνει η υπηρεσία σας σχετικά με αυτό. Επίσης, τι είναι με τα ελάχιστα κριτήρια προστασίας του περιβάλλοντος. Α, τώρα μπήκα στον πιασμό. να σας απαντήσω στα Ιταλικά. Τα Αγγλικά όμως. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ρωτάτε αφορά το πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον η εντολή της υπηρεσίας μας που θα έχουμε και περιβαλλοντικές ε, αρμοδιότητες. Σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό το, πρόγραμμα, το πρόβλημα. Δεν έχουμε ούτε νομική βάση ούτε εμπειρογνωμοσύνη. Δεν υπάρχει καν τέτοιο, τέτοιο πνεύμα, τέτοια κουλτούρα στην υπηρεσία μας. Πάντως προς τα εκεί θα κινηθούμε. Και γι' αυτό και σίγουρα χρειάζεται μια σαφής εντολή από Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα εντοπίσει το προβλήματα για το περιβάλλον σε σχέση με την ε, παραγωγή των φαρμάκων, σε σχέση με τα απόβλητα των φαρμακοβιομηχανιών. Πρόκειται για νέο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα, άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Θα δούμε ήδη τι έχει γίνει, οπότε θα πρέπει και εμείς έτσι να ε, εκπαιδεύσουμε υπαλλήλου για να ασχοληθούμε με το πρόβλημα. Οπότε ευχαρίστως και σε θεσμικό επίπεδο να αρχίσουμε αυτή την προβληματική για να δούμε πώς θα καλύψουμε και θα διεκπαιριώσουμε αυτά τα στοιχεία για το πώς θα πρέπει οι εταιρείε να υποβάλουν τα στοιχεία τους υπό άλλο σχήμα για να μπορούμε και εμείς να ασχοληθούμε με αυτό το πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει κάθε φορά να σκεπτόμαστε πέραν από την καλή πίστη που είναι σωστή αφετηρία τι γίνεται με τις επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους. Ο, όμως θα πρέπει να έχουμε και τους οικονομικούς πόρους σαν υπηρεσία. Συμπληρωματική συνομιλωσία Τι γίνεται με τα γενώσιμα και τα συναφή. Α, εδώ το πρόβλημα είναι λίγο πιο εύκολο. Ναι, θα πρέπει να διεκπαιρώσουμε το θέμα στη βάση της βιωσιμότητας όπως είπα στην αρχή της εισήγησής μου γιατί εδώ έχουμε δύο διαφορετικά θέματα. Πρώτα πρώτα την έγκριση αδειοδότηση εκεί που νομίζω ότι η αίμα και γενικά η Ένωση ε, μπορούν να προβούν στην έγκριση των δύο συναφών. Βρίσκομαι σε καλό επίπεδο. Όμως από την άλλη μεριά εδώ πέρα είναι δυσδιάκριτη η διαφορά όσον αφορά την εντολή που έχουμε. Γιατί το πολύ πολύ τι μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε κάποιες αντιθυντήριες γραμμές που θα αποφασίσουν και έτσι να προκαλέσουμε ανάληψη δράσης για να θα πρέπει να εγκρίνουμε ότι ήδη έχει τεθεί σε εμπορία. Μπορούμε να κλείσουμε τον πρώτο γύρο που είχε τις παρεμβάσεις των συντονιστών. Κλείνουμε με την κυρία Ντορνάνο από το ΕΝΕΦ. E σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ραζή. Θέλω να σας θέσω ορισμένα ερωτήματα. Μία από τις μεγάλες απειλές για τη δημόσια υγεία σήμερα είναι όπως ξέρετε η παραποίηση των φαρμάκων. Δεν μπορούμε παρά να φοβόμαστε λοιπόν ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των παραποιημένων φαρμάκων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ είναι το ερώτημά μου. Έχετε κάποιες προτάσεις σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές σε ό,τι αφορά τον αγώνα κατά των παραποιημένων <clears throat> φαρμάκων και σε ποιου θα μπορέσετε να στηριχτείτε για κάτι τέτοιο. Έχα ένα δεύτερο ερώτημα για τα γενώσιμα, αλλά έχετε απαντήσει ήδη και το τρίτο ερώτημα που είχα για την διαφάνεια στον φορέα σας. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη για την εξέλιξη του οργανογράμματος του φορέα σας και του προϋπολογισμού σας και τι συμπεράσματα θα εξαγάγετε στους επόμενους μήνες σχετικά με όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κέρια ερωτήματα, τα παραποιημένα φάρμακα. Έχουμε την οδηγία για τα φάρμακα μαϊμού, που είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το θέμα αυτό. Αλλά αυτό που με απασχολεί περισσότερο στον τομέα αυτό είναι η δυνατότητα αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ελπίδα μας είναι ότι με μια νέα παγκόσμια προσέγγιση, τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών θα μπορέσουμε και με την υποστήριξη της ε, Κομισιόν γιατί έχω απευθυνθεί ε, στο, στην Κομισιόν για το θέμα αυτό προσωπικά έχουμε πει ότι πρέπει να έλθουμε σε επαφή με τις χώρες όπου από προέρχεται το πρόβλημα αυτό κυρίως δηλαδή η Ινδία και η Κίνα Καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε μια ικανότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και το υποστηρίζουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά και η TTIP είναι ίσως ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη πεποίθηση. Πολλές φορές πηγαίνουν τρεις ή τέσσερις αρχές να επιθεωρήσουν το ίδιο εργαστήριο ή το ίδιο εργοστάσιο και αφήνουν άλλα χωρίς έλεγχο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια παγκόσμια δυνατότητα δημιουργίας ικανοτήτων για να ανακαλύπτουμε και να πατάζουμε τα παραποιημένα φάρμακα. Για την διαφάνεια και το οργανόγραμμά μας. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε σταθερή αύξηση των ανθρωπίνων πόρων στην αίμα. Ξέρουμε τώρα ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί βέβαια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον πρώτο γύρο οργάνωσης μπορέσαμε να έχουμε τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπίσουμε δύο σημαντικά νομοθετικά θεμάτα. Την φαρμακοεπαγρύπνηση και τις κλινικές δοκιμασίες. Τώρα ήδη μας ανησυχεί αυτή η αύξηση πολυπλοκότητος που θα προκύψει από τις νέες δραστηριότητε για να διατηρήσουμε ήδη την ποιότητα του έργου μας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το θέμα της ε, στελέχωσης του, του φορέα Ευχαριστώ που θέσατε αυτό το ερώτημα. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, κυρία Ντορνάνο. Όπως και εσείς και εγώ θα ήθελα να έχουμε την υποστήριξη Κομισιόν για τα παραποιημένα φάρμακα. Ναι, την έχουμε την υποστήριξη αυτή τον προηγούμενο μήνα. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ Στενάμε την Κομισιόν αποτελεσματικά. Και νομίζω ότι οι ρυθμιστές για τα θέματα αυτά έχουν υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση η οποία θα καρποφορήσει πολύ σύντομα γιατί είναι απαραίτητη. Thank you very much. now we can... Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε με τον δεύτερο γύρο, με την δεύτερη ομάδα. Ο Κρίστιαν Μπουζό είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ραζή, μετά από 20 χρόνια είναι επιτυχή η διαδρομή της ΕΜΑ στην Ευρώπη. Ήμουν μέρος της επίσημης αντιπροσωπείας. Συγγνώμη. Της ε, ΕΜΒ την Άνοιξη και παρά το γνώσο ότι δεν είναι και παρκώς τελεχωμένοι οργανίσεις, είμαι σίγουρος ότι με τη δική σας ηγεσία θα μπορέσετε να υλοποιήσετε τους στόχους σας. Όλες οι κλινικές δοκιμές που γίνονται στα παιδιά ε, στην ε, Ευρώπη, στις τρίτες χώρες καταγράφονται. Πιστεύετε ότι θα πρέπει η νομοθεσία να συμπεριλαμβάνει και τους ενήλικες ε, ε, οι οποίοι φύγανε αυτέ τι κλινικέ δοκιμές εντό και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεύτερη ερώτηση. Έχετε κατά νου πράκτικα μέτρα για να μπορέσει να αυξηθεί η συμμετοχή κρατών ε, εμπειρογνωμόνων κρατών μελών και κυρίως να έχετε και περισσότερους εθνικούς εκπροσώπους από τις νέες χώρες προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΕΜΑ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να έχω πολύ χρόνο για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Αν δεν σας πειράζει, αρχίζω από τη δεύτερη ερώτηση σας. Για την διεξιολόγηση των δραστηριοτήτων μας και τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις χώρες είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμεθα Έχουμε πολυεθνικές ομάδες, έχουμε τριπλασιάσει τον αριθμό των χωρών που ε, συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις ε, αξιολογήσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό και θα ενθαρρύνουμε τη συνέχιση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Η πρώτη ερώτηση. το θέμα της ε, καταγραφής όλων των ε, κλινικών δοκιμών που γίνεται και στους ενήλικες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προβλέψουμε. Με την FDA προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κλινικά ε, δεδομένα τα οποία έρχονται και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε, ε, αν είναι αξιόπιστα, πώς μπορούμε να τηρηθούμε σε τέτοιου είδους δεδομένα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και άλλες αρμόδιες αρχές. Εάν μια δοκιμή γίνεται εκτός Ευρώπης, αλλά τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται και στην Ευρώπη, θα πρέπει τα δεδομένα, τα σχετικά να τα έχουμε και σε μία βάση δεδομένων εντός Ευρώπης. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί η απάντηση. I'm Σας ευχαριστώ. Έκανα την ερώτηση αυτή διότι χιλιάδες ε, κλινικές ε, δοκιμές τέτοιου είδους γίνονται σε χώρες οι οποίες δεν έχουν ε, και πάρα πολλούς οικονομικούς πόρους και θα πρέπει να είμαστε ε, σίγουροι ότι ό,τι γίνεται και βάσει εθελοντών οι οποίοι συμμετέχουν σε δοκιμές ε, έχει αποτελέσματα τα οποία αν χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφαλή για τους πολίτες της Ευρώπης. Με την Επιτροπή ε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε ώστε να είναι πιο ελκυστικές δοκιμές ε, που γίνεται GCP, την GCP. Σας ευχαριστώ για την επισκεψή σας και αυτά που είπατε με τις απαντήσεις σας. Νομίζω ότι απαντώντας στο ερώτημα της κυρίας Ρης θέλω να μιλήσατε για την TTIP. Προφανώς αυτό δεν σας εμπλέκει άμεσα, αλλά θα ήθελα να έχω τη δική σας ε, εμπειρία και τη δική σας κρίση για το τι θα μπορούσε να προκύψει από μια ενδεχόμενη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την έγκριση φαρμάκων. Αν έχετε προβληματιστεί με το θέμα αυτό λοιπόν <clears throat> και επίσης σε σχέση με τις ε, ανάγκες των ε, ασθενών και όχι μονάχα από την οπτική γωνία της φαρμακευτικής βιομηχανίας ποια είναι τα ωφέλη που μπορούν να προέρχονται από τις τωρινές ε, συζητήσεις στα πλαίσια TTIP για τους ασθενείς και που είναι οι κίνδυνοι για τους ασθενείς. Δεν θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Δεν είμαι εμπειρογνώμων σε ό,τι αφορά τα εμπορικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν αυτό το οποίο μας ενδιαφέρουν και αυτό που είναι και αντικείμενο της προσπάθειάς μας και εδώ είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Κομισιόν και όλους αυτούς που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις της TTIP είναι να καταλάβουμε τις συνέπειες του τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι ότι δεν θα χρειαστεί να αλλάξουμε τις αρχές που διέπουν την διαφάνεια. Και για μας μια συνθήκη θα πρέπει να, για να γίνει δεκτή θα πρέπει να πείσει και την φαρμακοβιομηχανία για το κέρδος σε επίπεδο διαφάνειας που θα έχουμε με την πλήρη δημοσίευση των δεδομένων. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει πρόοδο σε επιστημονικό επίπεδο πολύ πιο γρήγορα με τον τρόπο αυτό. Και κατά δεύτερο λόγο, αυτά τα οποία είναι εμπορικό απόλυτο στην Ευρώπη είναι εμπορικό απόλυτο και αλλού. Το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα. Απλώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα τροποποιηθούν αυτά τα οποία κάνουμε ήδη και τα κάνουμε πολύ καλά και χωρίς προβλήματα. Επομένως, με ενδιαφέρει το να μην αλλάξουμε αυτά που έχουμε και σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συνέπειες δεν είμαι σε θέση να ξέρω. Είμαι εν αγνία του τελευταίου ε, προσχεδίου της ε, συνθήκης, επομένως δεν μπορώ να σας απαντήσω για το θέμα αυτό. Ίσως θα μπορούσα να μειώσω την άγνοιά μου. Όχι, δεν θέλετε συμπληρωματικό ερώτημα. Κύριε Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, κύριε Ράζη. Χαίρομαι ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία μα για τα θέματα τη υπηρεσία σα. Ε, έχω μια ερώτηση που δεν έχει ερωτηθεί προηγουμένω όσον αφορά την ε, χρήση των ε, φαρμάκων Εκτό. του IMM. Συνήθω, η αιτία είναι δημοσιονομική λόγη. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε κάποια εναλλακτική, κάποια διοδότηση από την υπηρεσία σας όπως δόθηκε άδεια στη Γαλλία να δοθεί ένα αντικαρκενικό φάρμακο σε κάποια ε, ασθένεια ή κάποια άλλη ασθένεια τέλος πάντων θα πρέπει η υπηρεσία να δώσει κάποιες καθημερινές γραμμές για τη χρήση φαρμάκων εκτός κατάλογο IMM. Για πέστε μας, πότε θα μπορέσετε να μας δώσετε αυτές τις κατευθυντήριες. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όσον αφορά τη χρήση αυτών των ε, φαρμάκων, αυτό είναι αιώνιο πρόβλημα, ξέρετε. Γιατί δεν υπάρχει φάρμακο τον οποίο να μην χρησιμοποιείται και σε κάτι το διαφορετικό από ό,τι προβλέπεται σε κάποια χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν ναι, συνέβαινε. Και με τη νέα, τις νέες κατευθύνσεις που υπάρχουν θα δούμε αυτό κατά πόσο ωφελεί και κατά πόσο είναι επικίνδυνο σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Και κατά πόσο επίσης μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Τώρα από πλευράς ε, ρυθμιστικής καθαρά ένα φαρμακευτικό προϊόν από τον νόμο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για σκοπό διαφορετικό του αρχικού μπορεί να οδηγήσει σε κάτι το επικίνδυνο. Είναι δυνατόν να γκρεμίσει το όλο οικοδόμημα της ρύθμισης. Βέβαια, αντιλαμβανόμεθα ότι στον πραγματικό κόσμο και με κάποια ρυθμική τεκμηρίωση δικαιολογείται μια τέτοια διαφορετική χρήση του προϊόντος του φαρμακευτικού οπότε και εμείς προσπαθούμε να ξέρουμε όσο γίνεται καλύτερα τι είναι ωφέλιμο και τι δεν είναι. Δεν είναι όμως εύκολο η υπηρεσία μας να μπορέσει να έχει όλα τα σχετικά στοιχεία γιατί πρόκειται για κάποια αυστηρή εντολή των εθνικών αρχών και οπότε εμείς θα πρέπει να μπούμε στα εθνικά χωράφια και βέβαια οι εθνικές υπηρεσίες δεν ενθουσιάζονται από τέτοια παρέμβαση ίσως σας απογοητεύει ότι δεν είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να, να σας δώσουμε το πλήρες τοπίο της ε, κατάστασης. Ίσως θα πρέπει κάτι να θεσμοθετηθεί ούτως ώστε να μπορέσουμε να το εντοπίζουμε το πρόβλημα. Ναι, αλλά για αυτή την περιπτώση μπορείτε να δώσετε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ. Επίση, μια δεύτερη ερώτηση. σας ανέφερα πριν για την διαφάνεια όσον αφορά τα τεστ, τα κλινικά, όσον αφορά τα όρφανα, φάρμακα, εσείς, πώς και έφτασε ότι μπορούμε να έχουμε την εξασφάλιση της ε, ανωνυμίας, ούτω ώστε αυτοί οι λίγοι ε, ασθενείς των σπανιών ασθενειών να μην επισημένονται. Γιατί τώρα έχουμε την υποχρέωση της πλήρους δημοσιοποίησης των στοιχείων για αυτές τις ε, κλινικές δοκιμές. Ράζει. Ναι, σας ευχαριστώ. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εμείς πασχίζουμε να δούμε τι θα κάνουμε για τη διαφάνεια των δεδομένων και την προστασία αυτών. Πρόκειται για μια από τις αιτίες για τις οποίες έχουμε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Γιατί όπως σωστά είπατε, πρόκειται για έναν περιορισμό που έχουμε πρόκειται για ένα όριο διαχωριστική κόκκινη γραμμή που δεν θέλουμε να την περάσουμε ούτως ώστε να μπούμε στα χωράφια του ιδιωτικού βίου. Οπότε και πιστεύουμε ότι τελικά θα λυθεί από τεχνολογικής πλευράς το πρόβλημα. Δηλαδή η τεχνολογία θα μας οδηγήσει σε κάποια λύση για το πώς θα μπορούμε να δημοσιοποιούμε τα σημαντικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επιστήμη χωρίς να εκθέτουμε και τα προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό και μέχρι τώρα έχουμε καθυστερήσει ε, κάποιες δημοσίευσεις γιατί ακόμα δεν έχει εξευρεθεί η λύση. Να, μια λύση όμως θα μπορούσε να ήταν η εξή. Να εμπλακεί και ο ασθενής. Εάν θέλει και προσφέρεται να συμμετάσχει στη δοκιμή στο πείραμα, ε, τότε θα θέλει και να δημοσιευθούν τα σχετικά δεδομένα του. Και θα μπορούσε αυτό βέβαια να καλύψει την πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι όλε Να μία πιθανή λύση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω που είστε εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων όπω, και συγγητή τη ομάδα μου και μένα η αηφορία των υγειονομικών συστημάτων και η πρόσβαση ε, στις ε, ναι, με απασχολεί. Ξέρω ότι εσεί έχετε ρόλο για να μπορέσετε να διασφαλίσετε την ασφάλεια των νέων φαρμάκων που κυκλοφορούν. Η αρχή τη ποιότητα ε, που πρέπει να ισχύει όταν δίδεται η έγκριση διαφόρων φαρμάκων πιστεύω ότι είναι κλειδί ώστε να μπορέσουν τα διάφορα κράτη-μέλη που είναι τα υπεύθυνα για τον καθορισμό των τιμών να έχουν την ασφάλεια. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο και η ερώτησή μου είναι ποιο είναι το πραγματικό κόστος της έρευνας, στο περίπου ίσως αν θέλετε, ποια θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στι ε, κλινικέ δοκιμέ, ώστε να δούμε πραγματικά ποια είναι η προστέμενη αξία τη ε, καινοτομία και να μπορέσουμε με ισοσκελισμένο τρόπο να καθορίσουμε τις τιμέ εκ μέρου των κρατών μελών. Επίση, κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σα για τι ε, αλλαγέ που γίνονται στην καινοτομία και επιτρέπουν στα σημερινά συστήματα που υπάρχουν για τα διάφορα φάρμακα ναι, ναι, ξέρουμε, κυρίως όσον αφορά τις ε, σπάνιες ασθένειες. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να δημιουργήσουμε κίνητρα ώστε να ενταθεί περαιτέρω η έρευνα κυρίως για τις σπάνιες ασθένειες. Thank you. It's a very question, <laughs> but... Um, το κόστος της έρευνας. Βασικά είναι το κόστος των κλινικών δοκιμών. Αυτό είναι το κόστος συν το κόστος της διάθεσης στο εμπόριο, το λανσάρισμα των νέων φαρμάκων. Στην... Ε, αυτό και είναι ένα μέρος της δικής μας εντολής. Θα πρέπει να δούμε με πώς μπορούμε και με την βελτίωση των συσκευασιών, με άλλα διάφορα θέματα μπορούμε να ελέγξουμε να έχουμε ε, πιο προσιτά οικονομικά φάρμακα αν θέλετε. Επίσης, σε πολιτικό επίπεδο θέλουμε βοήθεια. Εμείς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος και το περιθώριο κέρδους και ίσως μπορούμε να μειώσουμε το κόστος της έρευνας, αλλά κάποιος πρέπει να υποφεληθεί από αυτό το περιθώριο κέρδους που κερδίζεται. Δεύτερη ερώτηση. Good thing. Once again, there should be... Στη δεύτερη ερώτησή σας θα πω. Θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό που να μας επιτρέπει να μην έχουμε μόνο αύξηση του κόστους, αλλά και ε, κάποια κέρδη. Πολλές φορές όμως αυτό μας ξεπερνάει. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε εμείς ε, είναι να δούμε πού υπάρχει σε κάτι που γίνεται προστέμενη γινεται προσθεμενη ώστε να το ενισχύσουμε. Τώρα, ξέρουμε ότι τα φάρμακα για τις σπάνιες ασθένειες, τα ορφανά τα φάρμακα έχουν πάρα πολύ υψηλό κόστος και προσπά... γίνεται προσπάθεια από κάποιους να ε, παρέμβουν τις συνήθεις διαδικασίες και την νομοθεσία ώστε κάποια φάρμακα και κάποιες ασθένειες να συνεχίσουν να θεωρούνται ως σπάνιες, ίσως να προσθεθούν κι άλλες. Η κυρία Καβεσόν θέλει να προσθέσει. Όχι, όχι, νομίζω ότι ε, τον ε, χρόνο μου τον ε, εξάντλησα όλο. Μη Γαρδίνη. Yes. You change the order. <laughs> okay. Ε, σκουζάτε. Αχ, συμπαθάτε με λέει κύριε Γκραντίνη. Allora, io... Θα μπορούσα να είμαι πάρα πολύ γρήγορη, διότι πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα εδώ. Για να δούμε για να υπενθυμίσω αυτά τα οποία ήδη έχουν διηγηθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, όσον αφορά αυτό το οποίο είναι γνωστό ω ε, φάρμακα μαϊμού και παραπημένα και απομιμήσει. έχουμε κέντρα επιθεώρηση και έχουμε και στην Ευρώπη και έχουμε και στα τη μελη Αυτά επαρκούν ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεχής εποπτεία όσον αφορά την ποιότητα των φαρμάκων και ε, ε, αυτό το, το, το καινούριο σύστημα επιστοποίηση, ε, πανεπιστήμια κλπ. είναι δυνατόν να οδηγήσει σε επέκταση και διεύρυνση αυτού του ελέγχου και της εποπτείας των φαρμάκων. Τώρα τι γίνεται με τις προχωρημένες θεραπείες. Μας είπατε και μας είπατε για αυτήν την ε, ε, σχετική επιτροπή. Τι γίνεται όμως για αυτά τα οποία κάθε χρόνο εγκρίνεται. Νομίζω ότι οι εγκρίσεις είναι λίγες. Και όσον αφορά ε, όλη αυτή τη, τη δαπάνη που θα πρέπει να κάνετε για να συνεχίζετε η ζωή αυτής της επιτροπής από της ΕΜΑ για να έρχονται όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες δεν θα πρέπει κάτι να γίνει όσον αφορά την ε, Επιτροπή την άλλη που έχετε δεν θα μπορούσατε να συνδυάσετε το δουλειά των περισσότερων επιτροπών που έχετε τόσο ώστε να κάνετε κάποια εξοικονόμηση δαπανών τα φάρμακα από μιμήσεις βασικά έχουν σε δύο κατηγορίες πρώτα πρώτα αυτά που υπάρχονται στην εντολή μας δηλαδή, αυτά ε, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία GSP και GMP. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Ε, το κάνουμε και μπορούμε να το κάνουμε και ακόμα παραπάνω, να τα ελέγχουμε δηλαδή και να τα υποπτεύουμε. Και έτσι να μπορούμε να δράσουμε στην Ευρώπη. Όμως χρειαζόμαστε περισσότερους υπάλληλους επιθεωρητές. Ήδη έχουμε ένα κέντρο κατάρτισης στην Ευρώπη για αυτούς τους επιθεωρητάς. Και έτσι θα επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας και ε, η ωφέλεια θα είναι τεράστια για τις χώρες εκείνες όπου θα υπάρχει αύξηση επιθεωρητών. Σε δεύτερο επίπεδο τώρα. Σε επίπεδο εφαρμογής της νομοθεσίας. Αυτό είναι θέμα των διοικητικών αρχών της κάθε κυβέρνησης. Σε κάποιες χώρες οι διοικητικές αρχές είναι πολύ αποτελεσματικές στο να κάνουν τον έλεγχο αυτό σε επίπεδο χονδρικής, σε επίπεδο φαρμακείου και σε επίπεδο πελάτη. Άρα πρόκειται για αστυνομική δραστηριότητα. Αλλά επειδή έχετε βελτίωσει κατάσταση στην Ευρώπη, γιατί έχουμε κάποιε χώρε όπου υπάρχει λίγο ή καθόλου έλεγχο Τώρα για τι προκεχωρημένε θεραπείε. Ναι, λέτε ότι έχουν εγκριθεί πολύ λίγες, 5 ουσίε σε 10 χρόνια. Όμως ο, ο ρόλος των εμπειρογνώμων που είπατε είναι το λένε και πιο σημαντικός. Και εγώ είχα κάποιες επιφυλάξεις για την ε, αποτελεσματικότητα της Επιτροπής. Αυτή η Επιτροπή δεν είναι τόσο πολύ δάπανη, γιατί πρέπει να τη δείτε σαν επένδυση. Για πρώτη φορά διπλασιάσαμε σε ένα χρόνο τον αριθμό των επιστημονικών συμβούλων για τις προκεχωρημένες θεραπείες. Αυτό τι πάει να πει ότι για πρώτη φορά αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να δουλέψει όσο γίνεται πιο εντατικά. Και εν κατακλείδη να σας πω το εξής. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να γίνει συγχώνευση των δύο επιτροπών συγχώνευση και όχι κατάργηση της μιας εκ των δύο. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχετε συμπληρωματικό ερώτημα. Κύριε Αγκαντίνη, όχι. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσάλντες. Καλημέρα σας. Θέλω να μιλήσω για τις κλινικές έρευνες, την ηλικία και το φίλος ένα από τα στοιχεία της γυριατρικής στρατηγικής που ξεκίνησε από την ΕΜΑ το 2011 ήταν να εξασφαλιστεί ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούν οι πιο ηλικιωμένοι είναι υψηλή ποιότητα και δοκιμάζονται σε ηλικιωμένους το εγκριθούν. <clears throat> Μπορείτε να μας πείτε αν υπήρξε αύξηση της συμμετοχής των ηλικιωμένων σε κλινικές μελέτες νέων φαρμάκων και αν αυτό έχει βοηθήσει την αξιολόγηση αυτών των φαρμάκων για τους ε, ηλικιωμένου που έχουν διάφορες ασθένειες που οδηγούν στη λήψη φαρμάκων. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά αυτή η πολιτική. Επίσης, η ανισότητα σε σχέση με τα φύλλα στην κλινική έρευνα είναι κάτι που γίνεται και στο ζωικό βασίλειο γιατί χρησιμοποιείται και εκεί κυρίως ασθενικά ζώα. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι θα έχουμε μια σωστή γνώση των ε, επιπτώσεων των φαρμάκων όταν χρησιμοποιούνται μονάχα και δοκιμάζονται στο μισό πληθυσμό. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις κύριες ανησυχίες μας όταν αναλύουμε και αξιολογούμε τα δεδομένα. Για την γυριατρική. Πολλά έχουμε να κάνουμε ακόμα. η συμμετοχή των ηλικιωμένων ασθενών αυξάνεται, την προωθεί η Κομισιόν και υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις σχετικά. Αυτό το οποίο ελείπει ακόμα και με απασχολεί περισσότερο είναι ότι σήμερα δεν έχουμε τις επιστημονικές γνώσεις και τα υποδείγματα που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε το κύριο πρόβλημα της ηλικία. Δεν είναι τόσο η αλλαγή του μεταβολισμού, η αλλαγή στη δοσολογία, αλλά η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε άλλους παράγοντες στους οποίους εκτίθενται οι ηλικιωμένοι. Δεν έχουμε το επιστημονικό εργαλείο για να καταλάβουμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα φάρμακα σε ένα περιβάλλον πολυφαρμακίας. Έχουμε κάνει συζητήσεις για τα θέματα αυτά, αλλά δεν μας έχουν οδηγήσει σε σαφείς λύσεις. Ίσως χρειάζεται μια διαφορετική διαδικασία σχεδιασμού για τα φάρμακα και επίσης για τα δύο φύλλα. Ελπίζω και θα πω το ίδιο το οποίο είπα για τη γυριατρική και για τα δύο φύλλα. Για, με κάποιες ε, διαφοροποιήσεις γιατί για τα δύο φύλλα μπορεί να υπάρχει τελείως διαφορετική ε, αντίδραση στο διαφάρμακο λόγω του ορμονικού πλαισίου. Σε διαφορετικές ηλικίε υπάρχουν διαφορετικές ε, ε, αντιδράσεις. Αυτό το οποίο πιστεύω θα μπορούσε να το τμήμα της απάντησης είναι η έννοια των προσωπικοποιημένων φαρμάκων. Γιατί με την ε, αγορά φαρμάκων να είναι πιο προσαρμοσμένε σε βιολογικά προϊόντα, θα μπορέσουμε ίσως να θεωρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε ως υποομάδες το φύλλο και την ηλικία. Σας ευχαριστώ όλη κυρία Τσάρλες. Ελπίζω ότι σε, καμιά, σε πέντε χρόνια θα μπορείτε να πείτε κάτι περισσότερο από το ότι απλώς έχουμε ελπίδα. Γιατί εξαρτώνται οι ζωές πολλών ανθρώπων και όχι μονάχα οι ζωές των ανθρώπων. Αλλά η ποιότητα των ζώων των ηλικιωμένων εξαρτάται στην πρόοδο η οποία πρέπει να γίνει στην έρευνα και αν θέλουμε να έχουμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και περισσότερο, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει ειδική αντιμετώπιση για τις ηλικίε των ηλικιωμένων. Επομένως θα πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα και αυτό δεν θα συμβεί εάν δεν κάνουμε τις απαραίτητες προσπάθειες και το ίδιο με τις γυναίκες. Πάρα πολλές γυναίκες πεθαίνουν από καρδιακές, ε, καρδιοαγιακές ασθένειες και αυτό είναι υπερβολικό, είναι περισσότερο από ό,τι πρέπει να συμβαίνει. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι, εγώ είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Και επίσης θέλω να τονίσω ότι εμείς εστιάζουμε την προσέγγιση μας για την χρήση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπερχρησιμοποιούμε ορισμένα φάρμακα που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην εγκυμοσύνη και υποχρησιμοποιούμε άλλα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται λόγω της αγνίας και του ασθενούς και του ε, θεράποντος ιατρού. Επομένως και αυτό είναι ένα θέμα του προβλήματος. Ελπίζω θα μπορέσουμε στα επόμενα πέντε χρόνια να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ίσως και πιο πριν. Thank you very much. And now we can go to the next question, uh, Pilar Ayuso. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε και καλώς ορίσατε κύριε Ραζή. Αναφερθήκατε πολλές φορές στην φαρμακοεπαγρύπνηση το θέμα αυτό με ενδιαφέρει διότι ήμουν εισηγήτρια σκιώδες για τις, ε, ε, στις προηγούμενες θητείες για το θέμα αυτό. Σε σχέση με το θέμα αυτό πιστεύω ότι η ΕΜΑ έχει σχεδιάσει να επιταχύνει την έγκριση κάποιων φαρμάκων μέσω του Adaptive Pathways. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε αυτό. Και συμφωνείτε ότι αυτό είναι κάτι που θα δημιουργήσει αβεβαιότητα όσον αφορά την ασφάλεια κάποιων φαρμάκων που θα εγκρίνονται με ταχύες διαδικασίες. Τώρα, όσον αφορά την επαγρύπνηση που γίνεται στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να ενισχυθεί όλη η διαδικασία. Πώς προβλέπετε εσείς να ενισχύσετε αυτό το θέμα της φαρμακοεπαγρύπνησης και να υποστηρίξετε όλες τις δραστηριότητες λαμβάνοντας το κρατη Ευχαριστώ. Πρόκειται για τα, ε, μία, ε, τις πιο σημαντικές απαντήσεις που θα δώσω τώρα. Είναι πιλωτική αυτή η Adaptive Pathway Approach που είπατε. Ώστε να έχουμε, να αυτή την προσέγγιση ώστε καινοτόμα φάρμακα να διατίθεται στα αγορά πιο γρήγορα. Αλλά ξέρουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί συμπληρωματική αβεβαιότητα και ίσως κίνδυνος λέγουν κάποιοι. Αυτό όμως δεν ε, αληθεύει διότι λαμβάνουμε τα μέτρα μας και εκτός από την παραδοσιακή προσέγγιση Το ωφέλη θα είναι μεγαλύτερα αν δίδεται αυτή η επιταχυνμένη έγκριση. Διότι θα είμαστε πιο εστιασμένοι σε φάρμακα τα οποία θα διατίθεται. Τώρα, όσον αφορά την φαρμακοεπαγρύπνηση, είναι πολύ σημαντικό να είναι καλύτερη αυτή η επαγρύπνηση σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε, για να είμαστε αποτελεσματικοί, τις καλύτερο σχεδιασμό και καλύτερα αποτελέσματα. Όλες οι κλινικές μελέτες δεν μπορούν εκ των προτέρων να μας δώσουν όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας και με τον τρόπο αυτό θα είμαστε σε καλύτερη θέση εμείς ώστε να υπάρχουν καλύτερες και πιο ακριβείς απαντήσεις που θα δίδανται σε ε, περιπτώσεις ε, που τέτοιου είδους ε, φάρμακα δίδονται στην αγορά. Πιστεύετε λοιπόν εσείς ότι με τα μέτρα που διαθέτουν αυτή τη στιγμή οι διάφορες εθνικές ε, αρχές των κρατών μελών μπορούν ε, να επομισθούν αυτό το ε, συμπληρωματικό βάρος των εγκρίσεων. Όχι. Ναι. Πιστεύω ότι επαρκούν τα μέσα που διαθέτουν. Δεν χρησιμοποιούνται πλήρως και αν τα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε πλήρως θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί αν ενεργήσουμε όλοι από κοινού. Όπως σας είπα είναι πιλωτική αυτή η εφαρμογή και αν συνεχίσουμε θα, θα έχουμε τρεις εμπλεκόμενους που θα, είναι, ε, θα ενεργούν από κοινού. Τους ε, ασθενείς, τους ιατρούς και τους ε, υπεύθυνους των φαρμακοβιομηχανιών. Σας ευχαριστώ. Και για αυτό το τελευταίο τελευταία απάντηση. Τα τελευταία πέντε λεπτά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τις καταληκτικές σας παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου για την πολύ σωστά εστιασμένη ε, πολύ, πολύ εστιασμένες και συναρπαστικές σου ερωτήσεις. Έχω αντιμετωπίσει μόνο εν μέρη τα ερωτήματά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ και προσβλέπω στην δυνατότητα στο μέλλον να συζητήσω να είμαι ακόμα πιο σαφής και ακριβής και πιο εξαντλητικός και είμαι έτοιμος τα επόμενα πέντε χρόνια να δώσω όχι μονάχα απαντήσεις στα ερωτήματά σας αλλά λύσεις στα προβλήματα. Ξέρω ότι έχουμε μεγάλες προκλήσεις ενώπιών μας αλλά για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ευθυγράμμιση μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και έχω διαφορετική επαφή με την Κομισιόν. Υπάρχει κοινή συνειδητοποίηση των διακυβευμένων και είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ επικοδομητικός ο διάλογος που έχω με όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που έχουν δείξει μεγάλη υποστήριξη, ήταν πολλές φορές προκλητικά με επικοδομητικό τρόπο ή μας δώσανε και σημαντικές και καλές συμβουλές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much for your... Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, που ήρθατε εδώ. Γιατί ήταν εξαντλητική η κάλυψη των ερωτήσεων των συναδέλφων για σήμερα. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ και έχω να πω ότι το απόγευμα όχι, όχι το απόγευμα μόλις τελειώσει πρωινή συνδρίαση οι συντονιστές θα αποφασίσουν Οπότε και θα διαβιβάσουμε την απόφασή μας ή στον πρόεδρο κοινοβουλίου κατά την συνήθεια διαδικασία. Και τώρα. Α, τελειώσαμε πριν την προβλεπόμενη ώρα, οπότε πριν ε, το επόμενο σημείο το οποίο αφορά την ανταλλαγή απόψεων με τον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΚΑ ας περιμένουμε να έρθει σε ένα 20 λεπτό. Οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα για ένα καφεδάκι. Σύντομο διάλειμμα και 11.30 ξαναρχίζουμε. Θα τα πούμε σε λίγο.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 AUTHORWAVE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

καλή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 ο να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 δεν μόνο εγώ,

Υπότιτλοι Μελίδη Ουδάρη, πάρα πολύ φορτωτό, το σιωπηλό, κάθαμε με τον κόσμο που είχαμε, σε βάση Υπότιτλοι Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, και τώρα μπορούμε επιτέλους να αρχίσουμε. Έχουμε οργανώσει την ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Νταν Σέτ, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντή της ΕΚΑ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Χημικών Ουσιών και θα του δώσω <clears throat> το λόγο στον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΚΑ για να μας παρουσιάσει τις δραστηριότητες του φορέα του και θα αρχίσει η συζήτηση με απαντήσεις και μετά ερωτήσεις. Σας δίνω μέσα στο λόγο για την, ε, τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Με μεγάλη χαρά είμαι και πάλι μαζί σας για να έχουμε αυτή την ετήσια ανταλλαγή απόψεων. Στα επόμενα 10 λεπτά θέλω να κάνω τρία πράγματα. Πρώτα να παρουσιάσω τη γενικότερη εικόνα και να δείξω την πρόοδο που επιτυγχάνουμε προς την ε, εκπλήρωση της υποχρέωσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες. Στη συνέχεια θα μιλήσω πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα θετικά στοιχεία του REACH τα, τους καρπούς του ρίτς όπως τα έλεγα και τέλος θέλω να σας δώσω ένα ενσταντανέ για το που βρισκόμαστε στην εφαρμογή αυτής της ρηξικέλευτης νομοθεσίας. Το 2002 στο Johannesburg οι χώρες των Ηνωμένων Εθνών ήταν παρούσες στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορφής για την αϊφόρα ανάπτυξη και ένας από τους στόχους που δεσμεύτηκαν να πετύχουν ήταν μέχρι το 2020 χημικές ουσίες θα παράγονται και θα χρησιμοποιούνται με τρόπους που δεν βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην Ευρώπη προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου και ο κύριος μοχλός για αυτό είναι το REACH. Η χρήση και παραγωγή των χημικών ουσιών φυσικά είναι ευθύνη της βιομηχανίας, αλλά το REACH μας δίνει τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να διαδραματίσουμε το δικό μας ρόλο. Το REACH <clears throat> από τι εταιρείε να καταγράφουν και να θέτουν σε μητρό τι χημικέ ουσίε του και να περιγράφουν τα αποτελέσματά του για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Με αυτέ τι γνώσει, οι εταιρείε μπορούν να κάνουν καλύτερε και πιο ασφαλεί επιλογέ. Και εμεί τα κρατη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να κάνουμε τι απαραίτητε ενέργειε για να ελέγξουμε κινδύνους οι οποίοι θεωρούνται απαράδεκτοι για τους ανθρώπους και το περιβάλλον μερικά αριθμητικά στοιχεία για να δείξω την πρόοδο που έχουμε πετύχει για να φτάσουμε σε αυτό το συνολικό στόχο. 163 ουσίε υψηλή ανησυχία υπάρχουν τώρα στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να πετύχουμε να αυξήσουμε τον κατάλογο αυτό. 31 από αυτέ τι ουσίε απαιτούν πρόορη έγκριση, προ, προ, προηγούμενη έγκριση για να χρησιμοποιηθούν και μέχρι στιγμή 10 τέτοιε εγκρίσει έχουν δοθεί από την Κομισιόν και άλλε 60 γνωμοδοτήσει για άλλε αιτήσει έχουν δημοσιευτεί. Αυτές οι εγκρίσει δίνουν σε εταιρείε χρόνο να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις ενώ διατηρούν αυτές τις αγορές που έχουν και τις αλυσίδες προμηθειάς τους. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν λιγότερες αιτήσει για έγκριση από ό,τι περιμέναμε καταρχήν. Και πράγματι για μισές από τις <clears throat> ουσίες σε αυτόν τον κατάλογο έγκρισης δεν έχουμε δεχτεί καμία αίτηση. Πολλές από τις ε, εγκρίσεις είναι για παραγωγικές διαδικασίες και όχι για τελικά προϊόντα. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές δεν εκτίθενται σε αυτά τα προϊόντα. Παραδείγματο χάρη, το... η επικάλυψη στις βρύσες μπορεί να ε, ε, χρησιμοποιεί το τριοξίδιο του χρωμίου. Αλλά αυτό το οξίδιο χρησιμοποιείται μόνο στην παραγωγή της επικάλυψης που οποία είναι λαμπερή στις ε, βρύσες και όχι στο τελικό προϊόν. Επομένως μόνο οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτίθενται σε αυτό και εκεί υπάρχει η ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων. Είδαμε λοιπόν πολύ καλή διαχείριση κινδύνου σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα. Είμαι λοιπόν ε, σίγουρος ότι η διαδικασία της ε, εξάλληψης των πιο επικίνδυνων ουσιών συνεχίζεται <clears throat> και μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον συνολικό στόχο ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικές ουσίες. Σε μια στιγμή που τίθεται αμφιβόλο η νομοθεσία για το περιβάλλον σε όλο τον κόσμο και πολλές φορές ανατρέπεται, τώρα δουλεύει έχει αντίκτυπο και έχει θετικά αποτελέσματα τα οποία είναι απτά και ορατά. Δεν πρέπει βέβαια να επαναπαυόμαστε. Για πολλούς από εμά η εξάλληψη των πιο επικίνδυνων ουσιών δεν γίνεται αρκετά γρήγορα. Του χρόνου λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε την πρόοδο προς την κατεύθυνση των στόχων της ε, δέσμευσής μας για αηφόρο ανάπτυξη το 2020. Σε μια κίνηση συζήτηση με την Κομισιόν και τα κατημέλη θέλουμε να εντοπίσουμε τους τομείς όπου πρέπει να τροποποιήσουμε την εστίασή μας για να έχουμε καλύτερο αντίκτυπο. Προετοιμάσουμε την πενταετή μας <clears throat> αναθεώρηση της λειτουργίας του REACH, η οποία θα εμφανιστεί και στην αναθεώρηση της Κομισιόν το 2017 και συνολικά συλλογικά θέλουμε να κάνουμε το REACH να δουλεύει ακόμα καλύτερα και εγώ χαίρομαι για την ευκαιρία να συμμεριστώ τα συμπεράσματα αυτού του εργαστηρίου μαζί σας. <clears throat> και πάλι θα ήθελα να καταγραφεί η ευγνωμοσύνη μου για τη μεγάλη υποστήριξη που έχει λάβει η ΕΚΑ τα τελευταία χρόνια από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και από την, το σύνδεσμό μας την Julie Gerling. Το REACH είναι πράγματι μια συλλογική προσπάθεια. Πιστεύω ότι έχουμε καταδείξει την δυνατότητά μας να συνεργαζόμαστε από κοινού για να το κάνουμε μια επιτυχία το ΕΚΑ, τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Έμβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι πιστοποιημένοι συνομιλητέ και εμπλεκόμενοι και οι χιλιάδες εταιριών που <clears throat> συμμορφώνονται με το ΡΙΤΣ. Και τώρα, να προχωρήσω στα ωφέλη τα οποία μπορούν να προέλθουν από το ΡΙΤΣ και το πώ θα τα χρησιμοποιήσουμε. Όπω είπαμε προηγουμένω. το ΡΙΤΣ οδήγησε σε μαζική αλλαγή. Αλλά... Αντιστροφή του βάρου απόδειξη και έτσι ε, απαιτείται οι εταιρείε να ε, μοιράζονται αυτά τα δεδομένα. Υπάρχει καλύτερη διαχείριση του κινδύνου, καλύτερη επικοινωνία προ τα πάνω και προ τα κάτω στην αλυσίδα τη προσφορά και όλα αυτά είναι τεράστια αλλαγή όσον αφορά τη βάση δεδομένων. Και όλε αυτέ οι αλλαγέ απέδωσαν καρπού. Σήμερα όμω α επικεντρωθούμε στο τελευταίο από αυτά, δηλαδή ε, την βάση δεδομένων την Ιντερνετική online. Να σας δείξω κάτι. Πρόκειται για αυτή την κάρτα postal. Αυτή την κάρτα και σε παρακαλώ πάρτε μία πριν φύγετε στο, κοντά στην είσοδο στο βάθος της αίθουσας γιατί αυτό είναι απόδειξη αυτής της αλλαγής η οποία πιστεύω ότι πρόκειται να φέρει μία επανάσταση στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για τις χημικές ουσίες. Πιο απλά αυτό το Ιντερνετική βάση δεδομένων τώρα μας δίνει επιστημονικά δεδομένα σε 120.000 χημικές ουσίες. Και αυτές οι πληροφορίες τώρα υπάρχουν στο Ιντερνετ δωρεάν για όποιον θέλει να τα διαβάσει και να τα χρησιμοποιήσει. Και αυτό αφορά κάθε ουσία. Και υπάρχει επίσης και μια σύνοψη των επιστημονικών μελετών για τις επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον. Είναι η πιο μεγάλη βάση δεδομένων τέτοιου είδους στον κόσμο. Και κάθε μέρα βελτιώνεται και μεγαλώνει. Οι δε εταιρείε τώρα ε, υποβάλλουν νέε αιτήσει ε, καταχώρηση και ενημερώνουν τι καταχώρησει που υπάρχουν και αυτό είναι απίστευτα χρήσιμο για τους πανεπιστημιακούς, τις εταιρείες και όλους αυτούς που ασχολούνται με την ε, ασφάλεια των χημικών παντού και επίσης ε, χρησιμοποιείται από όσους ενδιαφέρονται για τις ουσίες και για τα αποτελέσματά τους, αλλά μόνο από αυτή, μόνο για αυτούς τέλος πάντων που έχουν αρκετή επιστημονική γνώση γιατί για όσους από εμά δεν τα γνωρίζουν δεν ωφελούν και πάρα πολύ οπότε γι' αυτό θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες για αυτή την ε, βάση δεδομένων με αυτή την επανάσταση Νομίζω ότι φέρνουμε μεγάλες αλλαγές και έχουμε τρεις κατηγορίες όσον αφορά το πολύπλοκο και έτσι νομίζω ότι θα αγγίξουμε ακόμη περισσότερο κόσμο. Στο πρώτο επίπεδο αυτό το οποίο το, εννοούμε, το, λέμε info card και αυτό μπορείτε να το δείτε σε αυτή την καρτούλα που σας είπα. Εκεί έχουμε τα βασικά. Πρόκειται για τις πληροφορίες που ωφελούν εσάς και εμένα, τους εργαζόμενους και τους προβληματισμένους καταναλωτές στο επόμενο επίπεδο υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες Ει δε το τρίτο και τελευταίο επίπεδο οι επιστήμονες μπορούν να διαβάσουν για τη χημική ουσία ε, τα πάντα αυτά πάνε και στη βάση δεδομένων τη δική μα. τώρα γιατί όλα αυτά σας τα επισημαίνω διότι ε, αφού θα είναι πιο προσβάσιμα αυτά τα δεδομένα εμεί θα εκμεταλλευτούμε ε, τους πιο πολύτιμους καρπούς του ρίτσου, δηλαδή τα δεδομένα. Ε, και έτσι έχουμε μια σημαντική επένδυση από τις ε, βιομηχανίες μετάλλου και χημικών προϊόντων στην Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι συμφέρον όλων να το εκμεταλλευτούμε. Για σκεφτείτε πόσο αξίζει αυτό για την πανεπιστημιακή και την βιομηχανική έρευνα, για την καινοτομία στη βιομηχανία, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία των καταναλωμένων και για το πόσο αυτό βοηθάει την ασφαλή χρήση της αναπτυσσόμενης χώρας. Καταλαβαίνετε τι θησαυρό είναι αυτά. Επίσης, ε, όπως τα βλέπουμε, αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείε για να συμμορφωθούν με τις ευθύνες τους για το περιβάλλον, για την υγεία, θα βοηθήσουν κατασκευαστές, λιανοπολιτές, καταναλωτές, να χρησιμοποιούν τις ουσίες με ασφάλεια, να κάνουν επιλογές πιο ασφαλείς για όσα κατασκευάζουν, για όσα πουλάνε και αγοράζουν και αυτό πρόκειται να δημιουργήσει συζήτηση στην αγορά, ώστε να υπάρχουν φιλικά στο περιβάλλον χημικά και θα αμυφθούν οι εταιρείε που καινοτομούν. Οπότε και εσείς μπορεί να έχετε έναν ε, ρόλο σημαντικό σε αυτή την επανάσταση. Αν αναρωτηθείτε ε, τι νομοθεσία παραπέρα μπορούμε να έχουμε για προσέγγιση του περιβάλλοντο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τα δεδομένα που ήδη έχουμε για το ρίτσι, για αυτό το σκοπό. Ας πούμε νομοθετικές μεταβολές που έχουν σχέση με τη βελτίωση του νερού, της ατμόσφαιρας, την ασφάλεια, στην εργασία, την υγεία και οι αρχές να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις πληροφορίες για το ρίτσο, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν και άλλοι στόχοι της πολιτικής μας. Ε, αυτό ε, θα οφείλουσε πάρα πολύ να το κάναμε την ε, βιομηχανία αλλά και τις αρχές. Τώρα να σας δώσω μια σύντομη εικόνα του που βρισκόμαστε. Βέβαια αυτή η συνοπτική εικόνα σας δείχνει πολύ λίγα πράγματα αυτό το τοπίο. Ε, τέσσερα πράγματα διάλεξα να σας δείξω και να σας πω ε, τι θα κάνουμε για τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών, πώς θα βοηθήσουμε μικρότερες εταιρείες, πώς θα ελαχιστοποιήσουμε τις αναγκαίες δοκιμές για ουσίες και ζώα και επίσης για τα βιοκτώνα, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πρώτα-πρώτα για τις ουσίες που έχουν περισσότερη σημασία, ακριβώς όπως είπαμε προηγουμένως για τους στόχους του 2020. Κάναμε εδώ αυτή την ε, επιλογή να εστιάσουμε την προσοχή στις ουσίες που είναι πιο επικίνδυνες για υγεία και περιβάλλον. Χρησιμοποιούμε αυτή την κατευθυντήρια γραμμή για να επιλέξουμε το ποια θέματα θα ε, εξετάσουμε ενδελεχέστερα και με αυτή την, ε, σε αυτή τη βάση με τα κρατημέλη αποφασίζουμε τι μέτρα διαχείριση θα πάρουμε. Και όπως γνωρίζετε, η ποιότητα των δεδομένων είναι κάτι που μας προβλημάτισε στο παρελθόν. Όμως, ε, όσο περνάει ο καιρό, η ποιότητα ε, βελτιώνεται και άρα οι αποφάσεις μας έχουν βάσεις πιο στέρεες. Οπότε για αυτές τις ουσίες που έχουν την πιο μεγάλη σημασία παραμένουν ακόμα δύο πονοκέφαλοι. Η ε, ενδοκρινική και νανοδιακοπές. Διαταράκτες, διαταράκτες. Νανοδιαταράκτες και ενδοκρινικούς διαταράκτες. Και σας είπα ε, ότι αυτό το έχουμε κάθε χρόνο, γιατί θα, δεν χρειάζεται να σας τα πω ξανά. Γιατί είπαμε ότι αυτά τα οποία γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις δεν είναι αρκετά στοιχεία για να να κρίνουμε κατά πόσον ε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προϊόντα με ασφάλεια και πολλές από αυτές τις αποφάσεις απαιτούν περισσότερες πληροφορίες όπως συζητάνε όλοι και έχουμε 5% από τις αποφάσεις των ελέγχων για, την, ε, για το σύνομο αυτών των φαρμάκων που έχουν ε, υποστεί ε, ένδικα μέσα και προσφυγές εναντίον τους. Είπαμε ότι ήταν 40% όσον αφορά τους νανοδιαταράκτες, οπότε όταν έχουμε κάποια προσφυγή αναστέλλεται η απόφαση και αυτό σημαίνει ότι, ότι οι εταιρείε δεν δίνουν πληροφορίες και δεν μπορούμε να μάθουμε για τις επιπτώσεις των ανωδιαταρακτών. Οπότε σας επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε πέρσι ότι η σύντομη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμφωνήσει όσον αφορά την αναθεώρηση των ε, προσαρτημάτων του ΡΙΤΣ και έτσι θα αρθούν όλες οι νομικές αβεβαιότητες. Και για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ε, κάτι παρόμοιο ισχύει. Τώρα προσπαθούμε ε, να δούμε πώς θα βοηθούμε τις διατάξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ε, αλλά ε, θα πρέπει να υπάρχουν και ευρωπαϊκά ε, κριτήρια γιατί αυτές οι ουσίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τρίτον, θα πρέπει να δούμε τι ισχύει για τις μικρότερες εταιρείε. ξέρουμε ότι το REACH είναι κάτι το πάρα πολύ απαιτητικό και αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στις μικρότερες εταιρείε και γνωρίζουμε ότι η επόμενη προθεσμία για καταχώρηση το 18 και αυτό πρόκειται να καλύψει πολύ περισσότερες από τις 3.000 που επιτυχώς έχουν καταχωρηθεί μέχρι σήμερα. Οπότε, όπως οποιοδήποτε σύγχρονος ε, ρεαλιστής νομοθέτης, ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να ελαφρώσουμε αυτή τη διοικητική επιβάρυνση. Να έχουμε καινούργια εργαλεία πληροφορικής, φιλικά στο χρήστη, για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως ε, τη βιομηχανία των εθερίων ελαίων κλπ. Αυτό βέβαια δεν κάνει τόσο πιο εύκολο το ρίζ για τους μικρότερους αλλά έχουν όμως ε, υλικό, έχουν κάποια προβλεψιμότητα τόσο ώστε οι εταιρείε αυτές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις όσο μπορούν πιο εύκολα. Και έτσι σήμερα μέρα, 50 από τους συναδέλφους μου επισκέπτονται 40 μικρές εταιρείε σε 13 χώρες ούτως ώστε άμεσα να αποκτήσουν μια εμπειρία για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές οι ΜΜΕ. Άρα έτσι θα καταλάβουμε πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Κατά τρίτον, θα πρέπει τώρα να δούμε πώς θα έχουμε όσο γίνεται λιγότερα πειράματα σε ζώντα ζώα και θα πρέπει να δούμε τι εναλλακτικέ υπάρχουν για αυτά τα πειράματα, αυτές τις δοκιμές ε, και επίσης έχουμε ενθαρρυνθεί από τους εμπλεκόμενους και το διαμεσολαβητή για να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να ληφθούν αυτές οι εναλλακτικέ υπόψεις στην αρχή της διαδικασίας πριν υπάρχουν οι προτάσεις για τα πειράματα στα ζώα προς την υπηρεσία μας και θα προσπαθήσουμε περισσότερο το χρόνο με όλους τους εμπλεκόμενους για να έχουμε ε, υιοθέτηση των αρίστων πρακτικών, να θεωρούμε τις ε, εταιρείες να χρησιμοποιήσουν τις εναλλακτικέ και επίσης την ε, μεθοδολογία που λέγεται QSAR που έχει να κάνει με τον ΟΣΑ. Επίσης συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε το πώς μπορούμε να έχουμε νέες ε, άλλου, άλλου τύπου μεθόδους άσχετες με τα ζωντανά ζώα ούτω ώστε να το χρησιμοποιήσουν εταιρείε οι οποίες θα καταχωρηθούν ε, εν ώψη της καταληκτικής του 18. Τέλος, πέρσι σας είπα για τα βιοκτώνα ποιο είναι το πρόβλημα και νομίζω ότι σε όλα τα μέτωπα που μας απασχολούν σημειώνουμε πρόοδο και έχουμε περίπου 500 εταιρείε τώρα που βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο. Ούτω ώστε αυτές μπορούν να παράγουν και να προσφέρουν ε, διοκτώνα. Και επίσης έχουν γίνει 11 αιτήσει για πανευρωπαϊκή αδειοδότηση για να τεθούν αυτά τα προϊόντα σε εμπορία. Και ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την υποστήριξη γιατί δείχνετε κατανόηση στα θέματά μας και βέβαια έχουμε λιγότερο προσωπικό το 16 για να επεξεργαστούμε όλες αυτές τις αιτήσει που δεν τις περιμέναμε. Παρακαλώ συνεχίστε να μας βοηθάτε και να μας βοηθήσετε να έχουμε το προσωπικό να διεκπαιρεώσουμε όλες αυτές τις αιτήσει, κυρίως που έρχονται από ΜΜΕ. Οπότε χρειάζεται η βιομηχανία να διατηρήσει την εμπιστοσύνη της στο νέο σύστημα για τα βιοκτώνα. Εμπιστοσύνη για την ευρωπαϊκή έγκριση, άδεια και για το ότι μπορούν να μείνουν ζωντανές αυτές τις στην αγορά. Ευχαριστώ κύριοι βουλευτές, πρόεδρε, για αυτή την ευκαιρία μας δώσατε. Ελπίζω ότι σας ενημέρωσα και σας προβλημάτισα και επίσης ε, ευχαρίστω να τα, να τα λέμε συχνά εάν θεωρείτε ότι θα είναι χρήσιμο. Εν πάση περιπτώσει, με ένα τηλεφώνημα ή με ένα email μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Thank ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, γνωρίζετε, έχουμε εργαστεί και εμείς για το σχέδιο της ΕΚΑ και κατά τη διάρκεια της ε, κατάρτισης του προϋπολογισμού στα πλαίσια της Επιτροπής Προϋπολογισμού ζητήσαμε να υποστηριχθεί η οργανωσή σας, διότι όπως ξέρουμε χρειαζόσαστε περισσότερες θέσεις και πόρους για να ανταποκριθείτε στο έργο το σημαντικό το οποίο πρέπει να φέρετε σε πέρα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κυρία Τάνσετ. Πολλά ακούσαμε στην, στην παρουσίασή σας. Πολλά θέματα τα οποία θέλω να θίξω. Ένα-δυο μας θα αναφέρω τελικά. Το πρώτο η προθεσμία του 2018 και την ε, συνειδητοποίηση από τους ε, τελικούς δείκτες αυτών των οποίων σημαίνει αυτό το θέμα. Εσείς ε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται με τους τελικούς χρήστες, κυρίως με τις ΜΜΕ. Καταλαβαίνετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουν όταν εκπνεύσει αυτή η προθεσμία το 2018. Εγώ πρέπει να πω ότι από όσον βλέπω και στην εκλογική μου ε, ε, περιφέρεια η συνειδητοποίηση και η ενημέρωση από κάποιους ε, γίνεται αργά και θα πρέπει εμείς να δώσουμε ένα σαφέστατο μήνυμα στις μικρές κυρίες επιχειρήσεις ότι το 2018 και μετά θα πρέπει να τιμήσουν τις υποχρεώσεις και να ε, μπορέσουν να συμμορφωθούν με αυτά τα οποία πρεσβεύει η ΕΚΑ. Δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρίως, απλώς να τις καλύτερα. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφέρω κάτι σε σχέση με το HVAC. κατά πόσον θα προσθέσει τον φόρτο εργασίας που έχετε, διότι θα πρέπει να δείτε και τα ε, ποσοστά που υπάρχουν από το HVAC και στα τελικά προϊόντα. Άλλαξε πολύ ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε ίσως σε αυτό το θέμα και μπορείτε να μου δώσετε ε, κάποιες εξηγήσεις και να μας ενημερώσετε. Και μια πιο γενική ερώτηση για το TTIP. Όπως γνωρίζετε, το συζητούμε το θέμα αυτό σε όλες τις επιτροπές στο Κοινοβούλιο και το συζήτησαμε πολύ και τα τελευταία χρόνια. Ένα από τα κύρια θέματα είναι το θέμα της ευθυγράμμισης των ε, κανονισμών και στα χημικά προϊόντα. Ανακαλύψαμε ότι όταν, ότι όταν πήγαμε στην Ουάσιγκτον ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Δεν τα κάνει πάντα όλα καλύτερα η Ευρώπη, αλλά υπάρχουν όντως μεγάλες διαφορές. Μπορείτε να σχολιάσετε το επίπεδο διαβούλευσης ε, για αυτό το θέμα που είχε με και με τον οργανισμό σας για διαπραγματευτική ομάδα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι είστε κατά κάποιο τρόπο θεματοφύλακας των ε, φιλοδοξιών μας αν θέλετε μέσω του Ρίτς. Μιλήσατε με αυτούς ε, για αυτά τα θέματα της ευθυγράμμισης των κανονισμών, κανονισμών στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που γίνονται από την Ευρώπη με τους Αμερικανούς για το TTIP. Ευχαριστώ, ο πρόεδρος. Δεν ξέρω αν κάποια άλλα μέλη θέλουν να θέσουν ερωτήματα τώρα. Κυρία Γκρός Τέτ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε και διευθυντά για την ανταλλαγή αυτή απόψεων που έχουμε μαζί σας. Παρακολούθησα αυτά που είπατε και παρακολουθώ και το έργο το οποίο φέρετε σε πέρασα. Υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτηματικά για τα νανοσωματίδια και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που είναι κέρια θέματα για την Επιτροπή μας. Να επανέλθω τώρα στο, στην προθεσμία του 2018 για την ε, καταγραφή ουσιών που χρησιμοποιούνται σε μικρές ποσότητες και θέλω να σταθώ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που είναι η παραγωγή εσάνς των ε, εθερίων ελαίων που είναι πάρα πολύ στην εκλογική περιφέρεια. Πολλοί θεωρούσαν ότι η η εσάν τη λεβάντας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι χημικό προϊόν. Ανα... Κατάλαβαν όμως την ανάγκη να συμμορφωθούμε του ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι τους τελευταίους 18 μήνες οι εκπρόσωποι των ε, γεωργικών και των βιομηχανικών ενώσεων είχαν πολύ σημαντικές ανταλλαγές απόψεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε με τον φορέα σας και με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να έχουμε σημαντική πρόοδο. Οι διάφοροι εμπλοκόμενοι εξάλλου έχουν χαιρετήσει την δέσμευση του δικού σας φορέα για να συνεχίσει αυτός ο διάλογος. Δείξατε ότι έχετε θετικό και ανοιχτό πνεύμα ώστε να μπορέσει να βρεθεί ένα σωστό πλαίσιο για αυτό τον οικονομικό τομέα ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει σημαντικές ε, και θετικές ε, κανονιστικές ρυθμίσεις που ήταν υπερπολύπλοκες όμως για τους παραγωγούς. Χαίρομαι λοιπόν για την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι όλες αυτές οι εργασίες οδήγησαν σε αίσιο πέρας και ποια θα μπορούσε να είναι η επίπτωση αυτών των συμφωνιών σε άλλους ευρωπαϊκούς τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκροστέτ για τα θέματα των εσάνς που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό και για μένα είναι. Γιατί στην ε, εκλογική μου περιφέρεια έχουμε πολλούς παραγωγούς τέτοιων ε, εσάνς και άλλων ουσιών και ενδιαφέρομαι και εγώ στο για το θέμα αυτό και τώρα η κυρία Μέλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντανσέτ για την ε, ομιλία του και για το γενικά του φορέα του. Εγώ είμαι κάπως καινούργια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσως φανεί αφελής η ερώτησή μου. Με ενδιαφέρει λιγάκι να ξέρω πώς ακριβώς λειτουργείτε όταν θέλετε να εκτιμήσετε τις τοξικές ιδιότητες μιας ουσίας. Πώς θα το κάνετε αυτό, το κάνετε μαζί με επιστήμονες κάτι αντίστοιχο με αυτό <clears throat> που γίνεται για την ΕΦΣΑ, δηλαδή υπάρχουν επιτροπές οι οποίες κάνουν ε, μια επιστημονική συζήτηση, θα ήθελα να μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει στο δικό σας φορέα. Πώς καταλήγετε στα αποτελέσματα αυτά, αναλάζουν τα αποτελέσματα με το χρόνο, υπάρχουν επιστήμονες από τα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μας τα παρουσιάσετε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μπάλτσο. Ευχαριστώ. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι επιχειρήσεις που διαθέτουν βιοκτώνα, οι εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν βιοκτώνα, πρέπει να έχουν έγκριση, αδειοδότηση ή να χρησιμοποιούν ουσίες που να ε, συνάδουν με τις ε, Όσον αφορά τη χρήση του ιωδίου, είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολείται η IRG Task Force. Η παραγωγή δεν είναι μέλος, είναι αυτού του consortium. Έχουν τον φάκελο που αφορά το ιόδιο που μόνο αν αγοράσουν τις πληροφορίες από την IRG Task Force. Η IRG καθορίζει από μόνη της τα κριτήρια ε, αποδοχής κάποιων ουσιών και κατά την άποψή μου υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. Θα ήθελα να μου πείτε, για ένα προϊόν όπως το ιόδιο, που δεν παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμμετέχει κάποιος στην ε, ε, σύσταση του φακέλου που επιτρέπει τη χρήση του, πράγμα το οποίο δημιουργεί πρόβλημα οικονομικό και αδυναμία κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Ντάνσετ για να απαντήσει. Α, συγγνώμη. Καλύτερα ίσως να ακούσουμε και την Επιτροπή τον κύριο Μπέρεν για να σχολιάσει την παρουσίαση του κυρίου Ντάνσετ. Και μετά θα δώσουμε το λόγο στον διευθυντή της ΕΚΑ για να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπω και τα μέλη τη επιτροπή σα, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάνσετ για την παρουσίασή του και πρέπει να πω ότι σε γενικέ γραμμέ μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά από τα πράγματα που ειπε σω Ίσως υπάρχουν ένα-δύο θέματα για τα οποία θα ήθελα να αντιδράσω, να μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε Ανέφερε προηγουμένως τις αδειοδοτήσεις, τις εγκρίσεις. Συμφωνώ ότι για πολλές ουσίες που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό δεν έχουν υποβληθεί αιτήσει. Το παράδειγμα που ανέφερε με το τριοξίδιο του χρωμίου και άλλες ουσίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στα τελικά άρθρα ίσως είναι πιο προβληματική η κατάσταση από τη δική μας προοπτική. Δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί πολλές αιτήσει από εταιρείε που τις χρησιμοποιούν αυτή την ουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουν ότι έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με ε, εταιρείε των τρίτων χωρών που δεν χρειάζονται αυτή την έγκριση και τελικά τα προϊόντα, τα τελικά που παράγουν οι δικές μας εταιρείε μπορεί να εισαχθούν από τρίτες χώρες. Πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας έγραψαν και τόνισαν το γεγονός ότι για τέτοιου είδους ουσίες αυτό το οποίο ανησυχεί κυρίως την βιομηχανία είναι η διασφάλιση θέσεων απασχόλησης. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο δεν προέρχεται μόνο από την βιομηχανία αλλά και πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπω προαναφέρω. Συμφωνούμε επίση πλήρω με τον κύριο Ντάνσετ με την αξιολόγηση που έκανε όσον αφορά την ε, ε, χρησιμότητα της ε, καταχώρηση. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της ΡΙΤΣ και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και σε άλλες περιπτώσεις και όταν αυτό κρίνεται ότι είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος. Τώρα, σε σχέση με τις ε, νανοουσίες και όντως η Επιτροπή προετοιμάζει την έκθεση ακτιολόγησης ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουν να μπουν στους καταλόγους τους ζήτη όλες αυτές οι νανοουσίες και τα νανοσωματίδια. Δεν είναι εύκολο, πρέπει να σας πω ότι αυτή η μελέτη αξιολόγηση δεν ήταν εύκολη, διότι χρειάστηκε να βρούμε τη σοσκελισμένη ε, μέθοδο μεταξύ κόστους ε, και γνώσεων που πρέπει να έχουμε, πράγμα όμως το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρίως για τις μιμίες. Στο τέλος του παρόντος έτους θα τελειώσει αυτή η μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων και θα σας κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ακούσατε τις ε, ε, εξηγήσεις της συναδέλφου της Επιτροπής Υγείας για την ε, οριστικοποίηση των κριτηρίων που αφορούν αυτούς τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Στο μεταξύ διάστημα πιστεύω ότι μπορούμε, έχουμε εμπιστοσύνη ότι δεν θα παραγνωρίσει αυτές τις ουσίες το ΡΙΤΣ. Κάποιες από αυτές είναι, είναι ουσίες οι οποίες μας ε, ανησυχούν πάρα πολύ και είναι τοξικές ως ουσίες. Ακόμη και στα συστήματα αναπαραγωγής, πράγμα το οποίο μας κάνει να είμαστε πιο σοβαροί για τον κατάλογο στον οποίο θα καταχωρούν. Τώρα, είπε ο κύριος Ντάνσετ ότι πολλά ε, μέλη του οργανισμού του πηγαίνουν επί τόπου σε μικρές ε, και μεσές επιχειρήσεις για να βλέπουν τι γίνεται και ποιο, πώς εργάζονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και έμαθαν πάρα πολλά πράγματα οι συνάδελφοι, διότι έμαθαν επί τόπου πώς έχουν τα πράγματα, πώς λειτουργούν οι εταιρείε, πώς μπορούν να υποστηρίξουν τις εταιρείε για να συμμορφωθούν με την νομοθεσία. Και τελικά ενθαρρύνουμε πολύ την ε, για να κάνει οτιδήποτε μπορεί ώστε να μειωθούν οι δοκιμές στα ζώα, κυρίως τα ζώντα, και να έχουμε πληροφορίες για ε, προϊόντα και χημικές ουσίες που δεν ε, δοκιμάζονται στο ζώο. Επίσης, η κυρία Γκέρλικ έκανε μια ερώτηση για το TTIP. Μπορώ να της πω με βεβαιότητα ότι βρισκόμαστε σε πολύ στενή σχέση με την ΕΚΑ και πάντα συζητούμε τα θέματα τα οποία είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση στην TTIP. Σήμερα το πρωί είπα κάποιους συναδέλφους ποιες είναι οι εξελίξεις για την ταξινόμηση των ε, ουσιών αυτών εκ μέρους των ΗΠΑ. Πρέπει να επαναλάβω ότι όντες στα πλαίσια του TTIP είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τους συναδέλφους της ΕΚΟ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Ντάνσετ. Ε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την καταληκτική προθεσμία του 2018, κυρία Γκέρλινγκ, που ήταν το πρώτο σας ερώτημα. Αναφέρεστε στους ε, κατάντι χρήστες. Ένα από τα προβλήματα του Ρίτς είναι ότι οι μικρές εταιρείες δεν καταλαβαίνουν πλήρως το ρόλο τους. Νομίζουν ότι είναι κατάντι χρήστες, ενώ μπορεί να είναι συγχρόνως και εισαγωγής κάποιων ουσιών που απαιτούν καταγραφή στο Μητρό του Ρίτς. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγματι να προσπαθήσουμε να φτάσουμε όλο και όσο δυνατόν περισσότερους εισαγωγείς για να καταλάβουν και αυτοί το ρόλο τους και την ανάγκη να αποφασίσουν κατά πόσο θέλουν να συνεχίσουν να εισάγουν αυτές τις ουσίες και να τις καταγράψουν στο Μητρό ή αν θα θέλουν να σταματήσουν αυτές τις εισαγωγές. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι κατάντι χρήστες έχουν και άλλες υποχρεώσεις και άλλες ανησυχίες από αυτούς που βρίσκονται σε άλλο σημείο της αλυσίδος. Αν αγοράζουμε λοιπόν χημικές ουσίες σε μικρές ποσότητες, μπορεί αυτές οι χημικές ουσίες να μην είναι πια καταγεγραμμένες. Και με τον τρόπο αυτό θα χάσουν την ικανότητα να συνεχίσουν να παράγουν τα προϊόντα τους με την τωρινή διαδικασία. Και για το λόγο αυτό θα θέλαμε να ανοίξουμε περισσότερες ε, δυνατότητες για τους κατάντι χρήστε να ελέγξουν πλήρως ποιες είναι οι προθέσεις σε σχέση με την καταγραφή των προμηθευτών τους. Οι κατάντι χρήστε επίσης έχουν πολλές υποχρεώσεις για να δίδουν δελτία σε σχέση με τα στοιχεία των προϊόντων τους, με τα ε, εμπλεκόμενες ουσίες στα προϊόντα τους και αυτό είναι μια μορφή συνεργασίας που έχουμε με αυτούς τους καταντιχρήστες για να τους βοηθήσουμε να, ε, να καταρτήσουν τα καλύτερα δελτία ασφαλείας για τα μείγματα τα οποία παράγουν όταν έχουν όταν έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία για τις πρώτες ύλες που πρέπει να τα κάνουν στοιχεία ασφάλειας για τα μείγματα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η πρόσφατη δικαστική απόφαση που ανέστηλε, δεν ανέστηλε στην πραγματικότητα, αλλά υπήρξε μια ανέστηλε μια ερμηνεία, υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ κρατών μελών, κάποιες ομάδες κρατών μελών και άλλων κρατών μελών και της Κομισιόν <clears throat> σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να ερμηνευτεί το κατά πόσο το 0,1% επηρεάζει το σύνολο του προϊόντος ή μόνο τις συστατικές του ουσίες και αποφάσισε το δικαστήριο ότι η σωστή ερμηνεία είναι ότι επηρεάζει τα πάντα. Όλα τα στοιχεία ενός ε, προϊόντος και έτσι είναι σημαντική και η ο ρόλος του ρίτς και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν έχουμε επιβεβαιώσει ότι θα τροποποιήσουμε τις οδηγίες που δίδουμε για, με μια επιταχυμένη διαδικασία ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η δικαστική απόφαση θα εφαρμοστεί γιατί είχε αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και με την επικείμενη, στην επικείμενη συνάντηση με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε καλύτερα την ε, νέα αυτή ερμηνεία αυτού του άρθρου για το REACH. Και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αποτελεί μία υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τις αρχές εφαρμογής και να τους δώσουν τα απαραίτητα εργαλεία και την κατάλληλη πρόσβαση στα δεδομένα σε αυτούς εναπόκειται στα λιμάνια να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου για να εξασφαλίσουν μαζί με τους λιανοπολιτές κατά πόσο οι προμηθευτές είχαν τις απαραίτητες πληροφορίες, είχαν δώσει απαραίτητες πληροφορίες για το τι περιέχεται στο προϊόν αυτό και ότι δεν περιέχει κάποια ανισχυτικού χαρακτήρα ουσία που να ξεπερνάει το 0,1%. Και για το θέμα της CHIP επιβεβαίωσε ο συναδελφός μου από την Κομισιόν το ότι γίνονται τακτικές διαβουλεύσεις με τους Αμερικάνους φίλους μας. Απλώς εμείς δεν είμαστε τμήμα των διαπραγματεύσεων καθόλου, μα καθόλου και ουσιαστικά απλώς παρέχουμε την απάντηση σε ερωτήσεις και ανταποκρινόμαστε στις ιδέες και τις προτάσεις περαιτέρω συνεργασίας με τους Αμερικανούς φίλους και συνομιλητές μας. Μια συνεργασία που υπάρχει επί τη βάση του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ε, Environmental Protection Agency. Για το ερώτημα της κυρίας Γκροστέτ που έχει να κάνει με τους παραγωγούς Essence, εθερίων ΕΛΕΩΝ Εγώ την ευχαριστώ γιατί κατανοήσω ότι έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες τον τελευταίο καιρό ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι απαιτήσει για το REACH σε ό,τι αφορά την καταγραφή των εθερίων ελέων θα πρέπει να είναι κατανοητές από τους παραγωγούς και εμείς θα δώσουμε την απαραίτητη υποστήριξη για να υπάρχουν κατατομής κατευθυντήριες γραμμές ώστε να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να εφαρμόσουμε καλύτερα το στον τομέα αυτό των εθέριων, εθέριων ελαίων. Και εγώ προσωπικά ήμουν παρόν στην τελευταία στρογγυλή τράπεζα στην Γκράς πρόσφατα και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι καταλήξαμε σε μια ε, συμφωνία για το πώς αυτές οι ουσίες που έχουν πολύτιμη σύνθεση μπορούν να εντοπιστούν. Είναι η διαδικασία HVCV. Τα έχουμε καταγράψει αυτά και στην ιστοσελίδα μας. Και έχουμε δεσμευτεί να τα μεταφράσουμε όλα αυτά στις, χώρες, στις γλώσσες των χωρών που έχουν αντίστοιχες παραγωγές με αντίστοιχες υποχρεώσεις ώστε και αυτές να εκμεταλλευτούν το έργο το οποίο έχει γίνει στην Γαλλία, διότι τα έγραφα αυτά βέβαια, όπως ξέρετε, είναι στα γαλλικά. Συνεχίζεται λοιπόν το έργο στο τομέα αυτό για τα οικοτοξικά αποτελέσματα της χρήσης ορισμένων ουσιών. Προσπαθούμε να δούμε τι ακόμα πρέπει να γίνει. Ελπίζουμε ότι μέχρι την άνοιξη του χρόνου θα έχουν συλλεχθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε οι παραγωγοί να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες για το ρίτς με έναν τρόπο που είναι αναλογικός και έχουμε καταγράψει και τον αριθμό των φακέλων που θα πρέπει να τύχουν καταγραφής και έχουμε και μια καλύτερη ε, κατανόηση του έργου που πρέπει να κάνουμε. Για αυτά που είπε η κυρία Μέλερ και το πώς αντιμετωπίζουμε το πρακτικό έργο του να έχουμε μια μεθοδολογία η οποία παρακολουθεί την πρόοδο της επιστήμης απλώς ήθελα να πω και πάλι και να υπογραμμίσω ότι το ρίτς αναστρέφει το βάρος απόδειξης ώστε οι εταιρείε είναι αυτές οι οποίες βάσει του πρέπει να καταδείξουν ότι τα προϊόντα τους και οι ουσίες που χρησιμοποιούν είναι ασφαλείς. Επομένως πρέπει να παραθέσουμε τις απαραίτητες αντίστοιχες μελέτες ώστε να έχουμε τις πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των ουσιών που χρησιμοποιούνται. Οι πληροφορίες αυτές μετά υποβάλλονται στο φάκελο εγγραφής στα Μητρώα και εξετάζουμε εμείς μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης. Το ΡΙΤΣ λοιπόν προβλέπει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τουλάχιστον 5% από τις καταγραφές σε σχέση με την ποιότητα της πληροφορίας η οποία παρέχεται. Και όταν έχουμε επιλέξει ένα φάκελο για αξιολόγηση, κάνουμε μια αναθεώρηση όλων των στοιχείων, μια επιθέωση των στοιχείων του φακέλου, να δούμε αν η ποιότητά του είναι επαρκής και ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες ποιότητος για το ρίξ. Και αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εκρίνουμε μια απόφαση περί συμμόρφωσης και ζητούμε από αυτούς που θέλουν να καταγράψουν την ουσία αυτή περαιτέρω πληροφορίες και αυτό το σχέδιο απόφασης αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο ο οποίος πρέπει να μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Και σε αυτή την περίπτωση επίσης διαβιβάζεται στην Επιτροπή του κράτους μέλους εκεί όπου έχουμε κάποιους συμπρογνώμενους από τα κράτη-μέλη και αναθεωρούν αυτές τις αποφασιστά σχέδια αυτών. Και το σημαντικό εν προκειμένου είναι ότι εξέλιξη του τι θεωρείται αποδεκτό και παραδεκτό ως ε, πληροφορία υφίσταται ενημέρωση με αναθεώρηση των παραδειγμάτων του ΡΙΤΣ που το κάνει η Κομισιόν ή με αναθεώρηση των κατευθυντηρίων. Οπότε ε, εξηγείται στον ετούντα την καταχώρηση πώς λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες του. Οπότε σχετικά με αυτό. έχουμε σε τακτή επαφή με αυτούς που ξέρουν τις εξελίξεις για τις μεθόδους των δοκιμών και πειραμάτων. Και λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη της επιστήμης στα πλαίσια της απόφασης για έγκριση νέων μεθόδων πειραμάτων. Οπότε έτσι ε, μπορούμε να έχουμε ενδεχομένω την αντικατάσταση των ε, πειραμάτων με ζώα. Και γενικώ στην υπηρεσία μας αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις της επιστήμης γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας από τους τέσσερις στόχους και προτεραιότητες για το μέλλον. Τους στρατηγικούς στόχους. Οπότε αυτό πάει να πει ότι ε, ε, ένα κομμάτι της δουλειάς μας γίνεται σε συνεργασία με κομισιόν και κράτη-μέλη και έτσι και νομοθετικά και ρυθμιστικά καλύπτονται ε, όλες αυτές οι διαπιστώσεις που έχουν σχέση με την εξέλιξη επιστήμης. Τώρα, η άλλη ερώτηση του κύριου Βάλχορτ. Έχουμε τώρα την απάντησή σας για την βιοεπιστήμη. Για τα βιοκτώνα, για τα βιοκτώνα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση έχουμε τους κανονισμούς, ένας από τους τέσσερις κανονισμούς που δουλεύουμε. Καλύπτεται από διαφορετικά κονδύλια του προπολογισμού. Οπότε και εξασφαλίζουμε το ότι τα έσοδα από τα διοκτώνα χρησιμοποιούνται για τα διοκτώνα και για το ρίτσο. Οπότε είναι ξεχωριστό κομμάτι τη δουλειά μα αυτό για τα διοκτώνα Τώρα, για το ιόδιο και τα σχετικά δεδομένα. Από ό,τι γνωρίζω, πρόκειται για μια ουσίες όπου βρίσκεται να εξελίξει το πρόγραμμα θεώρηση. Αυτό σημαίνει πώς. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εταιρεία που είναι ο βασικός ετών για την καταχώρηση και για τη θέση εμπορία του ιωδίου. Και ο νέος κανονισμός ορίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι εγκαίρως θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτό το παράρτημα. Τώρα όσον αφορά ε, την, την, την κοινοποίηση των δεδομένων το αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ θα γίνει η κατανομή του κόστου και των δεδομένων στην αγορά. Γιατί μια, μια, ε, μια μεριά είναι αυτοί που έχουν τα δεδομένα και την άλλη εκείνοι που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ε, στα δεδομένα στην αγορά. Και ε, επίση εδώ εφαρμόζεται η αρχή τη αναλογικότητα και αποφυγή διακρίσεων. Ανάλογα κάνουμε για να παρέμβουμε όπου υπάρχει κάποια διαφορά και προστριβή και αν κάποιες εταιρείε δεν μπορούν να τα βρουν έρχονται σε εμά για να τους κάνουμε κάποια δίκαιη κατανομή του κόστους. Όποτε χρειάζεται, όποτε υπάρχει μια τέτοια διαφορά, εμείς παρέμβουμε Να, τώρα έχουμε για το ιόδιο μια τέτοια περίπτωση και θα το κοιτάξω και θα σας πω. Επίσης, μας είπατε και για το θέμα της τρέβλης του ανταγωνισμού. Η συμμόρφωση με το δίκαιο ανταγωνισμού δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Αλλά εάν κάποια εταιρεία θεωρεί ότι συντρέχει κάποια παραβίαση αυτών των διατάξεων, τότε θα πρέπει να στραφεί στα εθνικά δικαστήρια. Να προσφύγει εκεί, αλλά επίσης να έρθει σε επαφή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, εάν σχετική δαπάνη μπορεί να την καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Πρόεδρε, νομίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις σαφείς απαντήσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ. Την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με εσάς κύριε Διευθυντά της ΕΚΟ και σας ευχαριστούμε και πάλι διότι είσαστε διαθέσιμος και απαντήσατε και σε όλες τις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι και θα τα πούμε σήμερα το απόγευμα, θα συνεχίσουν οι εργασίες της Επιτροπής μας. Τώρα θα παραμείνουμε στην αίθουσα για την συνάντηση των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ.